morning. No hammer. No hammer. Yes, Καλημέρα σας. Should be a hammer. No hammer. So, uh... Okay, good morning. Dear colleagues. Good morning, everybody. May I have your attention, please? Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορείτε να με ακούσετε. Good morning. If you take your seats, please. I guess the mic is okay. Τα μικρόφωνα δουλεύουνε, δεν άψω όλα. Your attention. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Με τιμά αυτή η ευκαιρία που έχω να ξεκινήσω εγώ και να κήρυξω την έναρξη αυτής της Επιτροπής των Πολιτικών ε, Ελευθεριών για την τρέχουσα κατάσταση. Εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη αν δεν έχετε αντιρρήσεις. Και καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση. Η συνεδρίαση. Ξέρετε ότι, έκτακτη συνεδρίαση, ξέρετε ότι στις 4 Ιουλίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε ένα ψήφισμα σε σχέση με το ε, πρόγραμμα των ΗΠΑ για, την, ε, για τις παρακολουθήσεις και τις σοβαρές επιπτώσεις του. Θα ήθελα να ακολουθήσω τους συναδέλφους από την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών και τους λοιπούς συναδέλφους. Εμείς ε, όταν, φέραμε, όταν ήρθε το θέμα ενώπιον της σκέψης των Πρόεδρων ε, αποφασίσαμε, ήμασταν αποφασισμένοι μάλλον ήδη, να συνεργαστούμε ενεργά. Η Επιτροπή των Εξωτερικών Υποθέσεων, η Επιτροπή, των, ε, Επιτροπή ΙΝΤΑ του Διεθνούς Εμπορίου που είναι συναρμόδιες για τα θέματα αυτά των παρακολουθήσεων και βέβαια βουλευτές των Εθνικών Κοινοβουλίων ενδεχομένως που θα ήθελαν να αναλάβουν πρωτοβουλία για να ρίξουν φως στην κατάσταση και τις συνέπειές της στο, ως προς την παραβίαση ιδιωτικής σφαίρας της ε, ζωής των ε, πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Και μετά και με αυτά περνάω στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης που είναι η πρόταση για συζήτηση. Πρώτα λοιπόν θα σας προσφέρω κάποιες πληροφορίες ύστερα από τη συνεδρίες της των Προέδρων της 4ης Ιουλίου. Μετά θα δώσουμε την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων γενική και στη συνέχεια θα ζητήσω από τη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης και τη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να τοποθετηθούν για να αντιδράσουν στα σχόλια που ενδεχομένως διατυπωθούν και στη συνέχεια και το Συμβούλιο το Συμβούλιο σήμερα συζητεί, από ό,τι γνωρίζω, ακριβώς τα ίδια θέματα. για να υποδείξει κάποιες λύσεις και εμείς βέβαια για τις ακροάσεις που σκοπεύουμε να οργανώσουμε πριν από το Δεκέμβριο θα κάνουμε προτάσεις με την ολοκλήρωση των εργασιών. Όπως είπα, στις 4 Ιουλίου είχα την τιμή εγώ να ε, υποβάλω στη διάσκεψη των Προέδρων την πρόταση. Ως Πρόεδρος Επιτροπής ε, Πολιτικών Ελευθεριών ε, προσεκλήθηνα από τον Πρόεδρο Μάρτιν Σούλτς να αναλάβω την πρωτοβουλία για μια, για μια εξέταση του ζητήματος από την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών. Ομόφωνα, ομόφωνα υπογραμμίζω, εγκρίθηκε η πρότασή μου. Και έτσι λοιπόν δείξαμε πνεύμα συνεργασίας, το οποίο υποστηρίζουν και άλλες επιτροπές. Είχα την ευκαιρία για μια ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Μπρόκ, Υπουργό, ε, Πρόεδρο της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων, για το θέμα αυτό. Και ως εκ τούτου, με χαρά καλωσορίζω τον κύριο Σαλαφράγκα, την κυρία Γκόμες και την κυρία Νέιτς, εκπροσώπους της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. θα θεσπιστεί μια ομάδα έργου απαρτιζόμενη από εκπροσώπου των διαφόρων υπηρεσιών του Κοινοβουλίου και των επιτροπών των συναρμοδίων των διαφορετικών επιτροπών για να ετοιμάσει ένα πρόγραμμα εργασίας για την Εξεταστική Επιτροπή. Για δίποτε υπόδειξη από τις πολιτικές ομάδες για το, τα πρόσωπα που θα πατήσουν και την γραμματεία για το σχέδιο του προγράμματος των εργασιών για τεκμηρίωση, εισηγητές, σκιώδεις εισηγητές που μπορεί να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ε, έγγραφα εργασίας και από το Σεπτέμβριο, και βέβαια για τις ε, ακροάσεις, από το Σεπτέμβριο η εξεταστική της ε, ΛΥΜΠΕ θα επικεντρωθεί στις δημόσιες ακροάσεις. Μια πρώτη υπόδειξη αφορά τον εξής κατάλογο προσώπων ή αρχών. Πρώτον, εκπροσώπους από τις Αμερικανικές Αρχές, εκπροσώπους του Συμβουλίου της Επιτροπής και του Συμβουλίου, της Προεδρίας δηλαδή. Τρίτον, εκπροσώπους των κρατών μελών. Τέταρτον, τακτική ενημέρωση από τις ομάδες υπηρεχνομόνων διατλαντικής συνεργασίας και ε, έκτον ειδικού εμπειρογνώμονες ε, για θέματα πληροφορικής ε, και κυρίως μεταφοράς δεδομένων προς την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των Πολιτειών ή ισοδύναμα συστήματα. Έτσι λοιπόν για να ξεκινήσουμε την προετοιμασία όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικά προτείνουμε η πρώτη ακρόαση να είναι αφιερωμένη στο, ευρωπαϊκό, στο αμερικανικό πρόγραμμα και τις νομικές του επιπτώσεις για τη θεώρηση διαβατηρίων. θα προσπαθήσουμε να προσκαλέσουμε τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπροσώπους της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και ειδικού σε σχέση με θέματα προστασίας δεδομένων, θέωρησης διαβατηρίων. Θα έχουμε εκπροσώπους από την EPIC και την ACLU αμερικανικές οργανώσεις και ως εκ τούτου θα πρέπει η διερεύνηση της υπόθεσης να καταλήξει σε συστάσεις, προτάσεις που θα συνοψίζονται σε ένα σχέδιο εκθέσεως το οποίο θα υποβληθεί στην όλο μέλη πριν το τέλος του χρόνου μάλλον και θεωρούμε ότι πολύ μεγάλη σημασία θα έχει ο χρονισμός Θέλουμε να καταθέσουμε ορατά αποτελέσματα πριν από το πέρας της θητείας του Κοινοβουλίου. Αυτό σημαίνει ότι θα εργαστούμε σκληρά για να έχουμε ένα σχέδιο εκθέσεως προς να υποβληθεί στην Ολομέλεια μέχρι το τέλος του έτους. Και βέβαια θα έχουμε και από το τμήμα πολιτικής στο Policy Department εκπληρογνώμονες που θα μας ενημερώσουν. Περιμένουμε τρία υπομνήματα ενημερωτικά από αυτούς για τα εξής θέματα. Πρώτον, ενημέρωση για το Αμερικανικό δίκαιο σε σχέση με το πρόγραμμα αυτό και ενημέρωση για τα εθνικά δίκαια και συστήματα μαζικών παρακολουθήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, να δούμε αν υπάρχουν τέτοιου είδους προγράμματα, γιατί ακούγονται πολλά για τη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Γαλλία, ενδεικτικά. Αυτή είναι μια γενική εικόνα της ανάλυσης την οποία θα μπορούσαμε να, προβούμε, να, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από το Γραφείο Ενημέρωσης, το Policy Department. Και επίσης για τα τέλη Οκτωβρίου. Έχουμε μια συνάντηση στη Ουάσιγκτον προγραμματίσει ήδη. Εγώ πρότεινα λοιπόν αυτή η αποστολή να γίνει από κοινού με τα μέλη της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων. Το πρότεινα στο Ιδέσκεψη των Προέδρων. Γιατί και εκείνοι είχαν προγραμματίσει μια επίσκεψη στην ε, πρωτεύουσα των ΗΠΑ τον Οκτώβριο. Παράλληλα λοιπόν να γίνει μια κοινή αποστολή με την ΑΦΕΤ μετά την παρουσίαση αυτού του πρακτικού πλαισίου δραστηριοτήτων. Θα ήθελα να σας ε, αναφέρω κάποια σημεία για το τι μας ενδιαφέρει. Καταγραφή της πραγματικότητας, συλλογή πραγματικών ε, στοιχείων, δεδομένων, καταγραφή ευθυνών, διαρεύνηση δηλαδή υποτιθέμενων ε, ε, παρακολουθήσεων από τις Αμερικανικές αρχές αλλά και από τις Εθνικές αρχές ε, ζημία, αξιολόγηση κινδύνου συνεπειών αυτών των παρακολουθήσεων ως προς τα θεμελιώδη δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και ιδιαίτερα το σεβασμό του ιδιωτικού βίου, του τεκμηρίου του δικαιώματος για άσκηση ενδικών μέσων σε περίπτωση δίκης αποτελεσματικά. Όλα αυτά ανθρώπινα δικαιώματα και θεμελιώδη δικαιώματα εγγεγραμμένα στο χάρτη ανθρώπινων δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερον, προστασία των προσωπικών δεδομένων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και για Ευρωπαίους πολίτες έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με ιδιαίτερη εστίαση στην αποτελεσματικότητα του ευρωπαϊκού δικαίου σε σχέση με, την, ε, με τους μηχανισμούς. Τρίτον, ασφάλεια, στην, ε, ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων στην εποχή του ε, ψηφιακού νέφους. Τέταρτον, ε, χρησιμότητα αυτών των συστημάτων παρακολούθησης για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Τέταρτον, αξιολόγηση των αποφάσεων για τις μεταφορές κρατουμένων σε τρίτες χώρες τις λεγόμενες ασφαλούς, ασφαλείς λιμένες ε, για περαιτέρω εκδίκαση προσφορά ενδίκων βοηθημάτων και μέσα ε, απόκρισης υποδίκου έβδομον περαιτέρω μέτρα για την προστασία σε υψηλό επίπεδο των προσωπικών δεδομένων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα με την υιοθέτηση ενός συνόλου μέτρων, ενός μια δέσμης μέτρων εκτεταμένης για, όλο αυτό το, για όλη αυτή τη θητεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και βέβαια αποκατάσταση δικαιωμάτων ύστερα από αυτές τις προσβολές, τις ε, προσβολές στην ασφάλεια αποκατάσταση της ασφάλειας ε, της ε, ψηφιακής στα, θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί από ό,τι μαθαίνουμε αυτά τα συστήματα παρακολούθησης έχουν φτάσει μέχρι τις ε, αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Washington, στην αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Washington και άλλους, άλλα διπλωματικά κτίρια ή κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του του λεχθέντος θα θέλαμε τις δικές σας θέσεις και προτάσεις, κατευθύνσεις και υποδείξεις για την περαιτέρω δουλειά. Σας εξήγησα λοιπόν τι είπα στη διάσκεψη των Προέδρων. Τώρα ήρθε η ώρα να σας ακούσω. Τι έχετε να πείτε. Σε κοινό λοιπόν με τον κύριο Κοέγιο που έχει στήσει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ε, επισημάνω ότι εμείς δεν πρέπει να ξεκινήσουμε εκ του μηδενός. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι καινοφανές και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή, από το τίποτα. Αντίθετα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γνωρίζει πολύ καλά αυτή την κατάσταση. Το 2000 και 2001 είχαμε συστήσει μια ειδική επιτροπή για την περίπτωση εσελών. Και τότε η Επιτροπή μας απέδειξε ότι είχαμε, υπήρχε ένα δίκτυο αγγλόφωνων ε, χωρών, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένο Βασίλειο, που αντάλλασαν πληροφορίες και έκαναν κατασκοπία. Κατασκοπία στην Ευρώπη. Η Επιτροπή Εσελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου απέδειξε με μαρτυρίες ε, ε, ηθινών των ΗΠΑ και παλιών διευθυντών της CIA ότι η μηχανή κατασκοπίας των Ηνωμένων Πολιτειών μετά τον ψυχρό πόλεμο ε, πέρασε από στρατιωτικούς στόχους σε οικονομικούς στόχους και μας εξήγησαν γιατί κατασκόπευαν οικονομικά την Ευρώπη. Δεν το αρνήθηκαν, δεν το διέψευσαν. Οπότε έχουμε ένα σημείο αφετηρίας, δεν ξεκινούμε εκ του μηδενός τότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έδωσε συνέχεια στα πορίσματα της Επιτροπής Εσελών. Γιατί η δημοσίευση των πορισμάτων συνέπεσαν με τα, τις τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νέα Υόρκη το 2001. Οπότε, χάρη αλληλεγγύης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ε, κρίναμε πολιτικός άσκοπο να χρησιμοποιήσουμε όλες τις πληροφορίες και τα πραγματικά περιστατικά που είχαμε. Αλλά αυτά τα πραγματικά περιστατικά και εκείνες οι πληροφορίες θα πρέπει να αποτελέσουν βάση εργασίας ε, στην ανάλυση της υπόθεσης πρίσμα. Δηλαδή δεν έχουμε κάτι το καινούριο, δεν έχουμε κάτι το πρωτοφανές. Έχουμε κάτι πιο εξεζητημένο απλώς τότε το σύστημα εσελών επέτρεπε την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνομιλιών, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αποστολή φαξ, τηλέτυπο, ε, δέσμες ε, αρτεσενές, ε, υποβρύχια, δορυφόρους και μάλιστα κάθε μισή ώρα αναλύονταν ένα ε, εκατομμύρια πληροφορίες, δηλαδή 48 εκατομμύρια πληροφορίες τη μέρα. Και μιλούμε για το 2000-2001. Αρκεί να λάβει κανείς υπόψη τη ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας από το 2000 μέχρι το 2013 για να αντιληφθεί πόσο έχουν προχωρήσει οι δυνατότητες ε, συγκέντρωση και ανάλυση των πληροφοριών στο μεταξύ. Οπότε, με βάση αυτά που είπατε, καλό θα ήταν να ξαναρίξουμε μια ματιά στα πορίσματα της TDIP που είχαν δοθεί σε όλα τα μέλη και τις μελέτες που αποτέλεσαν τη βάση του έργου της Επιτροπής και τον να ρίξουμε μια ματιά και στα ψηφίσματα της Ολομέλειας. Και δεν ξέρω αν θα ήταν και σκόπιμο σε μία από τις δημόσιες ακροάσεις να επενθυμίσουμε τους βασικούς πρωταγωνιστές της Επιτροπής, τον εισηγητή Γκέραρτ Σμιτ και άλλους που μας βοήθησαν με τεχνικές πληροφορίες ε, στην περίπτωση εκείνη. Τέλος ήθελα να πω ότι αυτό που είναι εις βάρος μας είναι περισσότερο ο χρόνος. Ο χρόνος τρέχει εις βάρος μας. Γιατί ουσιαστικά πριν τις ερηνές διακοπές δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα και στην πράξη του Κοινοβούλου θα κλείσει του χρόνου το Μάρτιο. Οπότε ελάχιστο χρόνο έχουμε στη διάθεσή μας. Και ο κίνδυνος είναι να οργανώσουμε εμείς Ακροάσει επισκέψεις, αλλά να μην καταφέρουμε να διεκπαιρεώσουμε τη διαδικασία και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Οπότε, ε, ίσως δώσουμε την, ευκαι... την εντύπωση ότι χανόμαστε σε επικοινωνιακές προσπάθειες και δεν ε, φτάνουμε στην ουσία του προβλήματος. Πιστεύω ότι θα έχουμε την ευκαιρία να καταπολεμήσουμε και να αποσοβήσουμε αυτό το κίνδυνο. Μα φυσικά κύριε Κοέλιο, όπως είπατε κι εσείς, είναι σαφές ότι δεν ε, πρόκειται να προχωρήσει η έρευνά μας πριν τις θερινές διακοπές. Ουσιαστικά η πρόταση θα υποβληθεί αμέσως μετά το καλοκαίρι, αμέσως μετά τις θερινές διακοπές, 5 Σεπτεμβρίου, που θα έχουμε την ε, συνεδρίαση και θα προσπαθήσουμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο το Σεπτέμβριο, ώστε να αναπτύξουμε τη στρατηγική μας. Ο κύριος το λόγο. Um, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι γιατί ο κύριος Κοέλιο ξεκίνησε με το θέμα του έσυλον. Είναι όντως πολύ επικοδομητικά όλα αυτά και ο λόγος για τον οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό το παράδειγμα αυτό είναι γιατί ήταν μια άσκηση συλλογής ε, στοιχείων και ένα από τα, πρόγραμμα, τα προβλήματα της άσκησης αυτής ήταν ότι ξεκίνησε με κάποια κριτήρια τα οποία είχε θέσει η γραμματεία για, αυτήν, ε, για την περίπτωση αυτή που ήταν ε, η, η διαχείριση των προσδοκιών και η, η έρευνα των πηγών και τότε τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε με το Εσλόν ήταν ότι όταν αρχίσαμε να ε, συζητάμε και να μιλάμε με τους, ε, με, τα, ε, με τους υπευθύνους τέλος πάντων των υπηρεσιών πληροφοριών είχαμε, αντιμετωπίσαμε κάποια προβλήματα με τις κατασκοπίες και τα λοιπά. Εμείς σαν κοινοβούλιο είμαστε διατεθειμένοι υποτίθεται να συζητήσουμε κάποιες φήμες που κυκλοφορούν, κάποιες πληροφορίες που κυκλοφορούν και κάποιες πληροφορίες από αυτές αφορούν τους πολίτες, άρα πρέπει να αντιδράσουμε και πάρα πολύ καλά κάνουμε και αντιδούμε σαν ε, κοινοβούλιο, όμως ε, ε, θα είμαστε περιορισμένοι όπως και στο, και στο έσυλον. Άρα πρέπει να μπορούμε να διαχειριστούμε τις, ε, προσδοκί, τις προσδοκίες μας. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Ότι για τα πρώτα δύο κριτήρια τα οποία έθεσε η γραμματεία πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και διάφανοι απέναντι στους πολίτες μας και παρεπιπτόντος ο κατάλογος πρόεδρε τον οποίο ε, έχετε συντάξει για τις ε, ε, ακροάσεις ε, δεν συμπεριλαμβάνει την, ε, τις ITPS και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις πρέπει να τις συμπεριλάβουμε γιατί σε αυτές τις ακροάσεις πρέπει να είμαστε ανοιχτοί και όταν συγκεντρώνουμε πληροφορίες πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, πραγματιστές όσον αφορά την διαχείριση των πληροφοριών, των προσδοκιών μας διότι δεν θα φτάσουν ποτέ σε μας κάποιες πληροφορίες όπως και στο ΕΣΛΟΝ. και από την άλλη πλευρά υπάρχει και το χρονοδιάγραμμα που, έθεσε, το πρόβλημα που έθεσε ο κυρία Κοέλιο, ε, υπάρχουν τομείς που εμείς σαν κοινοβούλιο μπορούμε να προσφέρουμε κάτι παραπάνω. Για τα σημεία 4, 5 και 6 ε, που είναι η επανόρθωση, η δικαστική, η ε, νομική, ε, η κάλυψη των κενών κτλ. Εδώ η πρόκειται για πολύ σημαντικούς και πυκνούς αν θέλετε τομείς και αν είμαστε λογικοί και μεθοδικοί μπορούμε να μπούμε στην ουσία των προσδοκιών των πολιτών μας. Δεν θέλω ε, να, να, να, να, μιλήσω περισσότερο για να, και να πάρω τα, ε, τον χρόνο των συναδέλφων, αλλά όταν συζητάμε για τα διάφορα θέματα ε, στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τουλάχιστον, γιατί οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων θα μιλήσουν για τον εαυτό του, είχαμε πει ότι χρειαζόμαστε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων. Άρα έχουμε προλάβει, αν θέλετε, κάποιες από, τις, από τα θέματα τα οποία μας απασχολούν τώρα, π.χ. η μεταφορά των πληροφοριών. Εμείς θέλουμε να υπάρχει μια ρύθμιση όσον αφορά την μεταφορά των πληροφοριών ε, για εμπορικούς λόγους και να, υπάρχει, να, είναι πλαισιωμένη και η λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών. Λοιπόν, ε, η κατασκοπία, το να βρούμε πληροφορίες κτλ. είναι θέματα δύσκολα και δεν θα έχουμε πρόσβαση σε αυτά τα θέματα όπως και για το Έσυλον δεν είχαμε. Ο, τύπο, ο τύπος βέβαια θα μας παρακολουθεί από κοντά, γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε και προσεκτικοί για το πού θα βάλουμε τον πύχη των προσδοκιών μας όταν ξεκινήσουμε. Άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να δούμε τι το κοινοβούλιο, τι προσδοκίες μπορεί να ικανοποιήσει το κοινοβούλιο, διότι και με το SWIFT και το PNR πάλι στην ίδια κατάσταση ήμασταν και πρέπει να ικανοποιήσουμε τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πολιτών μας και να είμαστε θετικοί. Το σημειώσαμε. Η κυρία Βέμπερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για το, τις γενικές γραμμές και για το πλαίσιο της συζήτησης. Βέβαια οι αποφάσεις ε, θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασής μας. Τρία πολύ σύντομα σχόλια. Καταρχάς, οποιαδήποτε και αν είναι η πραγματικότητα, υπάρχει και η αντίληψη της πραγματικότητας. Και εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είμαστε υπεύθυνοι και για αυτή την αντίληψη της πραγματικότητας που έχουν. Γι' αυτό πιστεύω ότι το πιο, η πιο σημαντική πτυχή στις δραστηριότητες ε, στους επόμενους μήνες σε σχέση με το θέμα αυτό είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πλήρη διαφάνεια. Οτιδήποτε συζητήσουμε εδώ είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπορούμε να μοιραστούμε με τους Ευρωπαίους πολίτες. Η, αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα πολύ ισχυρό ε, μια πολύ ισχυρή τάση αν θέλετε στην, ε, στις πολίτες και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατά των, πολιτο, κατά των χωρών και των κυβερνήσεων γιατί ε, υπάρχουν φήμες που κυκλοφορούν ότι και κυβερνήσεις κρατών μελών ήταν εμπλεγμένες σε αυτές σε αυτού του είδους τα πράγματα. Άρα θα πρέπει την απέτηση που έχουν οι πολίτες να τη υπόψη μας και να δείξουμε ότι δεν έχουμε να κρύψουμε τίποτα ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα, ούτως ή άλλως ξέρουμε ότι θα ληφθεί μια πολιτική απόφαση. Το γνωρίζουμε αυτό. Όμως πρέπει στους πολίτες μας, το αξίζουν οι πολίτες μας να γνωρίζουν όλα τα γεγονότα και να τους εκθέσουμε ακριβώς τα γεγονότα. Ανεξάρτητα από το που έλαβαν χώρα τα γεγονότα αυτά, από τη μία από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Και επιμένω ότι στις ακροάσεις μας, και πραγματικά ειλικρινά τώρα μιλάω, δεν πιστεύω ότι αυτές οι δραστηριότητες με τις έρευνες κτλ. κτλ θα πρέπει να έχουν σαν τελικό σκοπό μία έκθεση μία έκθεση, μπορεί να καθίσει κάποιος σε ένα γραφείο ακόμα και τώρα και να την ε, συντάξει. Αυτό είναι σημαντικό, αυτό που είναι σημαντικό είναι να συλλέξουμε, να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν σε αυτήν την έκθεση. Γι' αυτό θα πρέπει να δούμε και τις δραστηριότητες των δικών μας κρατών μελών και όχι μόνο των εταίρων μας στις ΗΠΑ. Και ίσως να ήρθε ο καιρός, γιατί μια και μιλάμε ε, τόσο πολύ για τις συμφωνίες ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες και η αλήθεια είναι ότι για το PNR και για το SWIFT τους έδωσαν ό,τι μας ζητήσανε. Ίσως επομένως να ήρθε η ώρα να ξαναρχίσουμε την συζήτηση για την ε, προστασία των προσωπικών δεδομένων στα πλαίσια της συνεργασίας Ήπα Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην αρχή ήταν σημείο και μετά εξαφανίστηκε. Ευχαριστώ κυρία Βέμπερ. Ο κανονισμός για το πρόγραμμα Πρίσμα ε, ε, έχει σε φω σε αντίστοιχε πρακτικές που εφαρμόζουν και τα κράτη-μέλη εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε αυτή η έρευνα στη ΛΥΜΠΕ αφορά και αυτό το θέμα. Θα συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τους μηχανισμούς και τις δραστηριότητε του προγράμματο Πρίσμα, αλλά ταυτόχρονα και για τις πρακτικές των κρατών μελών σε ό,τι αφορά μαζικές παρακολουθήσεις. Ο κύριος Άλμπρεχτ τώρα, έχετε το λόγο. Thank you very much. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τους συναδέλφους που εγείρουν πολύ σημαντικά ζητήματα, ιδιαίτερα τον κύριο Κοέιο. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να ρίξουμε φως στα πραγματικά περιστατικά και τις προτάσεις που είχαν γίνει και συμφωνώ και με την Ρενάτη Βέμπερ ε, να ρίξουμε φως και να εξηγήσουμε στους πολίτες τι έχει συμβεί όπως τότε με την Επιτροπή Εσελών του κ. Κοέλιο. Είναι πολύ σημαντικό και στα κράτη μας να στραφούμε προς τις αρχές και να διατυπώσουμε τα ερωτήματα, διότι πρέπει να πω ότι περίμενα ήδη να έχουμε προσκεκλημένους κάποιους σήμερα από τις αρχές αυτές για να ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα αυτή την εξεταστική δουλειά. Γιατί ξέρετε βέβαια ότι όταν ο Guardian απεκάλυψε την, ε, το πρόγραμμα για τις φυλακές ε, το, το πρόγραμμα Πρίσμα ε, την επομένη ακριβώς ε, η Βουλή των Κοινοτήτων στο Ηνωμένο Βασίλειο άρχισε μια εξεταστική επιτροπή. Εμείς έχουμε αφήσει να περάσει στους καιρός και αρχίσουμε να συζητάμε τώρα πώς θα κάνουμε τη δουλειά. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να αφήσουμε να γελιοποιηθούμε. Ας ξεκινήσουμε την εξέταση, ας βάλουμε το πρόγραμμα μπρος, να δώσουμε μια ευκαιρία στους πολίτες να ενημερωθούν για το τι συμβαίνει και γι' αυτό καλώ τους πάντες να επιταχύνουμε το έργο, να μην ξεκινήσουμε στα τέλη Σεπτεμβρίου, αλλά μέσα μετά το καλοκαίρι. Να αρχίσει η διερεύνηση από την πρώτη συνεδρίαση και μαζί με τα Εθνικά Κοινοβούλια, γιατί πρέπει να τους προσκαλέσουμε το ταχύτερο δυνατόν να έρθουν, από τις εξεταστικές επιτροπές ε, για τις ε, μυστικές υπηρεσίες των Εθνικών Κοινοβουλίων που έχουν την αρμοδιότητα ως τέτοιες επιτροπές να διαρευνήσουν τη δράση των μυστικών τους υπηρεσιών γιατί πρέπει να μας ενημερώσουν να δούμε πώς ε, αντιλαμβάνονται τις αποκαλύψεις αυτές και ενδεχομένως συνδέσμους και σχέσεις μεταξύ των διαφόρων προγραμμάτων που υπάρχουν. Πρέπει να προσκληθεί και η Europol. Και ο κύριος Wainwright. Γιατί πρέπει να δούμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα όργανα της και οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες, εάν ήξεραν, εάν είχαν υπόψη τους και τι από όλα αυτά. και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ε, καλέσουμε και το Συμβούλιο και παρακαλώ να, μετα... μεταφερθεί στο Συμβούλιο το ε, μήνυμα ότι οι αρχές ε, οι εθνικές θα πρέπει να στείλουν αντιπροσώπους τους εδώ γιατί είμαστε το κατάλληλο μέρος για να θέσουμε τον δάκτυλο επί των τύπων των ύλων και μην ξεχνάμε ότι και αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων στην Ευρώπη δεν έχουν αναλάβει ακόμα, δεν έχουν λάβει ακόμα απαντήσεις, έχουν ζητήσει να γίνουν έρευνες και ε, ανακρίσεις για την εμπλοκή και των μυστικών υπηρεσιών. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να προσκαλέσουμε και εκείνους οι οποίοι έχουν ε, αποκαλύψει την αλήθεια όπως ο Edward Snowden, τους λεγόμενους whistleblowers. Είναι πολύ σημαντικό βέβαια να τον δούμε. Αλλά και άλλους, το Mark Klein από την AT&T, πρώην συνεργάτη της AT&T, ο οποίος είχε ανακαλύψει το μυστικό δωμάτιο ε, που είχε στόχο να εκτρέψει δεδομένα ε, backbone, ε, σπονδυλικά δηλαδή δεδομένα, αλλά και άλλους και πρώην προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών των ΗΠΑ και βέβαια και Ευρωπαίους whistleblowers όπως τους λέμε που έχουν αποκαλύψει τέτοιου είδους προγράμματα. Πολλοί επίσης ε, από το χώρο των πανεπιστημίων θα ήταν ενδιαφέρον να προσκληθούν ε, ο κύριος Κάσπερ Μπάουντεν και άλλοι που έχουν κάνει έρευνες και μελέτες για το λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήταν ένα παράδειγμα. Και βέβαια ο Γκέρτ Σμιτ, όπως είπε ο κύριος Κοέλιο, και άλλοι που θα ήταν χρήσιμο να προσκληθούν, αλλά δεν θα σας δώσω εκτενή κατάλογο τώρα των ονομάτων. Όπως είπα θα πρέπει να αρχίσουμε ήδη την διερεύνηση της υπόθεσης. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι έχουμε περιορισμένες αρμοδιότητες εδώ Δεν μπορούμε εμείς να επιβάλλουμε περιορισμό στη δράση των εθνικών υπηρεσιών, άλλωστε δεν είναι και ρόλος της Επιτροπής μας. Πρέπει όμως να εξετάσει το πώς αντιμετωπίζονται και οι παραβιάσεις αυτές του κράτους δικαίου και των συνθήκων. Αυτό θα πρέπει να είναι το αντικείμενο των συνεδριάσεων μας. Θα πρέπει να συζητήσουμε την... Ε, το συσχετισμό μεταξύ των εθνικών μέτρων σε σχέση με την προστασία της εθνικής ασφάλειας και της δικής μας θεώρησης, αν τα θέματα αυτά είναι όντως θέματα εθνικής ασφάλειας ή αν ε, υπάγονται στον χώρο των συνθήκων, στο πεδίο των συνθήκων, γιατί δεν πρέπει να αφήνουμε κενά και δεν θα πρέπει να επιτρέπουμε στα κράτη-μέλη να εκτρέπονται ε, από το σεβασμό των βασικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό λοιπόν πρέπει να κάνουμε και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Και πρέπει να το κάνουμε με πνεύμα ανοιχτό προ του πολίτε. Θα πρέπει να στραφούμε προ τα εθνικά κοινοβούλια και να δούμε και οι δικές τους αντίστοιχες εξεταστικές επιτροπές, γιατί αυτέ θα δραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο όταν έρθει η ώρα να κρίνουμε τι μυστικέ υπηρεσίε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Άλμπρεχτ. Σημειώνουμε όλε τι προτάσεις. Προσοχή συνεδρίαση τη εξεταστική μα επιτροπή, ήδη προβλέπεται για τι 5 Σεπτεμβρίου σα υπενθυμίζω. 5 Σεπτεμβρίου ώστε να ξεκινήσουμε το ταχύτερο δυνατό. Άρα θα γίνει η ίδια εξέταση τότε, θα έχουμε εξεταστικές διαδικασίες ανακριτικές. Ναι, στις 5 Σεπτεμβρίου και υπογραμμίζω και εγώ από πλευράς μου την σημασία της επικοινωνίας με τα εθνικά κοινοβούλια για να δούμε τα ίδια θέματα και τώρα ο κύριος Κίρκοπ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ξέρετε ότι υπάρχει μια ασθένεια που ονομάζεται ε, η τρέλα του μεσοκαλόκαιρου. Έχει και κλινικά χαρακτηριστικά βέβαια, αλλά κυρίως κοινοβουλευτικά σε τέτοια εποχή. Εγώ έχω πει ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι να καταγραφούν τα πραγματικά περιστατικά πρώτα πριν να ξεκινήσουμε τις ανακρίσεις και τις εξετάσεις. Διαφορετικά θα είναι πολύ γελία εικόνα που θα δώσουμε. Και η Επιτροπή, ξέρετε, το έχει άλλωστε πει ξεκάθαρα, έχει κληθεί να εξετάσει τα θέματα αυτά και να τεκμηριώσει ενδεχόμενες παραβιάσεις ελευθεριών, δικαιωμάτων και το καθεξής δυνάμει του δικαίου της Ένωσης και κυρίως των συνθήκων. Με ενδιαφέρον άκουσα τον κατάλογο των ε, πιθανών εντός αγωγικών μαρτύρων που επικαλείται ο κύριος Αλμπρέχτ. Συναρπαστικός κατάλογος. Εάν περιλάβουμε κάποιους από αυτούς που μας λέει, ελπίζω να είναι ακόμα όλοι στη ζωή, αλλά κάποιοι δυστυχώς ε, που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν έχουν ε, αποδημήσει κύριων. Ο Μάρκους Βόλφ, επί παραδείγματι, ε, θα ήταν πολύ χρησιμό, αλλά δυστυχώς έχει αποδημήσει. Ο κύριος Βλαντιμίρ Πούτιν, ε, αρχηγός της ΚΑΓΚΕΜΠΕ και της FS5 μεταξύ θα μπορούσαμε να δώσουμε κάποιες πληροφορίες για την ΚΑΓΚΕΜΠΕ που ήταν η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά τα χρόνια Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε και αν ακολουθήσουμε το δρόμο αυτόν. Ξέρουμε πολύ καλά ότι μπορούμε να απευθύνουμε ευγενικά μια πρόσκληση στους επικεφαλείς των μυστικών υπηρεσιών των διαφορών κρατών μελών για το G10, για το Πρίσμα και, το, και όποιο άλλο πρόγραμμα βεβαίως μπορούμε να, θέλουμε, να τους πούμε ότι θέλουμε να έρθουν να μας μιλήσουν αλλά φοβ... υποψιάζομαι ότι ενδέχεται να είναι κάπως απασχολημένοι και να μην βρούνε χρόνο γιατί ίσως να ασχολούνται με τίποτα κυβερνοεπιθέσεις και τρομοκρατίες. Εν πάση περιπτώσει όμως. Ναι, ναι, όντω ασχολούνται με πολλά θέματα, ξέρετε, προστατεύουν τα συμφερόντά μα ανά τον κόσμο. Δεν νομίζω λοιπόν αυτόν τον χρόνο να έρθουν. Και θα ήθελα να καθίσω σοφέ το εξή. Ότι πρώτον, αντιτίθεμαι ρητά σε οποιαδήποτε απόπειρα να προσκληθούν, να μας μιλήσουν οι οι κατηγορούνται για διάπραξη σοβαρών αδικημάτων. Η αναφορά στο όνομα του κυρίου Σνόουντεν ήταν τελείως άκερη. Δίνει τελείως εσφαλμένα μηνύματα σε οποιονδήποτε θα ήθελε στην Ευρώπη να διαλευκάνει την υπόθεση και δεν φανταζόμουν ότι θα μπορούσε η αδίποτε πολιτική ομάδα να εκφράσει τις θέσεις. Βεβαίως κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να, να... να βεβαιωθούμε ότι γίνονται σεβαστοί οι νόμοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ότι η αδίποτε παραβίαση αυτών ε, υποβάλλεται για εξέταση στις εθνικές αρχές, γιατί δεν νομίζω την αρμοδιότητα της Επιτροπής μας ή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εν όλο ε, η εξέταση αυτών των θεμάτων. Και έτσι, Πρόεδρε, για να βοηθήσω κι εγώ από πλευράς μου σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή θα έρχομαι ε, να, να κάνω κάποιες παρατηρήσεις. Αλλά εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε ως Επιτροπή τις ε, οργανώσεις, τους, φορούς, τους φορείς και τις υπηρεσίες αυτές που προστατεύουν τους πολίτες μας από εξωτερικούς ε, ή εσωτερικούς εχθρούς και που προστατεύουν τις δημοκρατίες, άσχετα με το πώς βλέπουν τη δημοκρατία ορισμένη εδώ μέσα. Σας ευχαριστώ. Όλα τα σημειώνουμε προσεκτικά. Και μην ξεχνάτε ότι ακολουθούμε εντολή της Ολομέλειας. Ήταν ψήφισμα που ενέκρινε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Εκεί έγινε η σύσταση για την Ερευνητική Επιτροπή, για την έρευνα αυτή που πρέπει να διεξαγάγουμε, με το σκεπτικό ότι ναι, μεν οι Ευρωπαίοι πολίτε ενδιαφέρονται για την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, αλλά ταυτόχρονα είναι γεγονό ότι ε, δεν είναι σίγουρο ότι τρομοκρατικέ επιθέσει ή απειλέ ε, θα εκπορευθούν από την Ευρωπαϊκή Πρεσβεία στις Ηνωμένες Πολιτείες ή από ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Ελάχιστη είναι η πιθανότητα να πλέκονται τέτοια σχέδια εδώ. Επίσης, οι διαπραγματευτές της συμφωνίας ε, με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, πρέπει να τα λάβουν αυτά υπόψη. Πέρα λοιπόν ε, αυτού του υπόβαθρου της, του αντιτρομοκρατικού αγώνα, έχει νόημα να γίνει αυτή η έρευνα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως ε, αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ανέθεσε το καθήκον σε εμά. Κυρία Ένστ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γιατί όχι το Βλάντιμιρ Πουτίν. Πολύ ενδιαφέρον θα ήταν. Αν και δεν είμαι σίγουρη ότι θα ερχόταν για τον κύριο Σνόντεν όπως και για τα υπόλοιπα ονόματα μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον ο κατόλογος που ακούστηκε κύριε Κέρκοπ. Αν πρόκειται πάντως για προσκλήσεις, νομίζω ότι θα πρέπει μέσα στην εβδομάδα παραδείγματι να δώσετε την ευκαιρία κύριε Πρόεδρε στις ομάδες να καταθέσουν προτάσεις για να μπορέσετε μετά να ξεχωρίσετε Είχαμε πέρσι ένα, μία έκθεση ε, για τις παρακολουθήσεις και την κατασκοπία ε, από το project για τις παρακολουθήσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να τους προσκαλέσουμε και αυτούς για να δούμε τι έχουν να πούνε. Θα έχουν πολλά να πούνε και ενδιαφέροντα αυτά ως προς τα πρόσωπα. Βέβαια το δίλημα. Το δούλημα μας είναι ότι δεν έχουμε την κλασική ανακριτική επιτροπή και κύριε Κύρκοπ, ναι πράγματι Ισχύει αυτό που είπατε, αλλά εγώ λυπούμε που δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να εξετάσουμε τα πραγματικά περιστατικά και ως εκ τούτου πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας σε αυτά που μπορούμε να κάνουμε. Ωστόσο, μη έχοντα την ανακριτική εξουσία, θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί αυτό με απασχολεί πολύ, αν μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τα ε, στοιχεία που χρειάζονται για να διερευνήσουμε την κατάσταση. Ξέρετε ότι εδώ πολύτιμα, πολύτιμα θα είναι τα τεκμήρια, τα ντοκουμέντα, τα έγγραφα δηλαδή που θα μπορούσαμε να συλλέξουμε και γι' αυτό θα ήθελα όσο δυνατόν περισσότερα έγγραφα να έρθουν στην προσοχή της Επιτροπής μας. Για το Έσυλον και τον κύριο Πουέρτας, Κοέλιο, συγγνώμη, ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε η εμπειρία από αυτή την Επιτροπή ποια ήταν, σε τι αποτελέσματα κατέληξε και θα έλεγα ότι ναι, χρειάζεται μια πραγματική ανάλυση. Όπως είπα, πολύ φοβούμαι ότι δεν θα έρθουν όλα τα έγγραφα, οι εμπειρογνώμονες που θα θέλαμε να δούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας προσπαθήσουμε και αν δεν καταφέρουμε μέχρι το πέρατος της θητείας να ε, δώσουμε ένα πραγματικό, μια πραγματική έκθεση για την υπόθεση αυτή, τότε νομίζω θα πρέπει να ομολογήσουμε μια τραγική αποτυχία. Γιατί αυτό περιμένουν οι πολίτες για να, ε, να αποκαλυφθεί η κατάσταση, αλλά βέβαια και οι επιχειρήσεις οι οποίες αντιλαμβάνονται ότι κοιμούνταν ήσυχα ενώ κάποιοι τις παρακολουθούσαν. Για να το πω έτσι. Και πρέπει πάνω απ' όλα να κοιτάξουμε το χρόνο. Χρειαζόμαστε μια παράλληλη με την ε, τακτική επιτροπή οργάνωση των συνεδριάσεων της εξεταστικής. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είναι μια κανονική επιτροπή που απλώς οργανώνει κάποια workshop. Όχι, χρειάζεται μια πραγματική στρατηγική που θα έχει το δικό της προγραμματισμό και πάνω απ' όλα πρέπει να στραφούμε στα εθνικά κοινοβούλια και να αφιερώσουμε φερρυπίν 14 ημέρες όπου θα ασχοληθούμε μόνο με την υπόθεση αυτή. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι δυνατόν ή νοητόν να ε, ακολουθήσουμε τον τακτικό ρυθμό των συνεδριάσεων μιας κοινοβουλευτικής επιτροπής. Χρειάζεται μια διαφορετική στρατηγική για την οργάνωση του χρόνου και των συνεδριάσεων και αυτή θα έχει τεράστια σημασία στο αποτέλεσμα. Και χρειάζεται και μια κοινοβουλευτική στρατηγική. Πώς θα το χειριστούμε το θέμα αυτό. Έχουμε ένα ψήφισμα στο οποίο λέμε ότι το PNR και το SWIFT πρέπει να, ε, να διακοπούν, να διακοπεί η λειτουργία τους. Τι κάνουμε λοιπόν, ε, προχωρούμε αμέριμνοι, ε, συνεχίζουμε με τις συμφωνίες για την ανταλλαγή πληροφοριών, την προστασία προσωπικών δεδομένων που ακόμα δεν υπάρχουν σε σχέση με τις ΗΠΑ, διακόπτουμε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Τι είδους στρατηγική λοιπόν ως κοινοβούλιο μπορούμε να προβάλλουμε, αυτό πρέπει να το συζητήσουμε και με σοβαρότητα διαφορετικά θα ξεφουσκώσει όλο αυτό σαν μια ε, φούσκα μεγάλη η οποία τρύπησε, χωρίς αποτελέσματα δηλαδή. Και ξέρετε ότι ο κόσμος, ο πολίτης δεν ενδιαφέρεται ούτε για το πόσες ώρες θα έχουμε συζητήσει εδώ, ούτε για το πόσα έγγραφα ή εμπειρογνώμονες θα έχουμε δει. Θέλει να δει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα και το αποτέλεσμα έχει τη μεγαλύτερη σημασία ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Γιατί τέτοιο είδους, τέτοιο είδους σκάνδαλο δεν έχουμε ξαναδεί στην ιστορία μας. Ευχαριστώ κύριο Μπρόγκ, έχετε το λόγο. Ήρθε η σειρά σα. Ευχαριστώ. Την περασμένη φορά μιλούσαμε για συγκέντρωση πληροφοριών, παρεμβατική συγκέντρωση από τις ΗΠΑ, αλλά με ανησυχεί περισσότερο για διάκριτη ε, χρήση και ανταλλαγή αυτών των πληροφοριών. Και ε, αυτή η έρευνα μπορεί να ξεκινήσει ε, ως έρευνα για σημαντικό, έρευνα για σημαντικό έγκλημα, αλλά μπορεί να καταλήξει σε συγκέντρωση που δεν έχει κλιματικό χαρακτήρα ή συγκέντρωση προ, προσωπικών πληροφοριών για άλλους λόγους. Το 2011-2012 η συγκεντρωση προσωπικων πληροφοριων για αλλους λογους το 2011 2012 η κυβερνηση των ΗΠΑ προσπάθησε να νομοθετήσει για θέματα τηλεφωνικών ε, συνομιλιών ε, ή ε, στοιχείων για ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αλλά δεν ευωδόθηκε αυτή η νομοθετική απόπειρα. Τώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο για γνωστούς λόγους και κυρίως για την προσωπική ελευθερία δεν ψήφισε αυτή τη σχετική νομοθεσία και τελικά αποφάσισε ότι δεν χρειαζόταν τη χειροποθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου γιατί έπαιρνε τις πληροφορίες αυτές και πολύ περισσότερες από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Βίλιαμ Χέιγκ, ο Υπουργός Εξωτερικών, του ε, ε, ερωτήθηκε για το θέμα αυτό από το Κοινοβούλιο και δεν το διέψευσε κατηγορηματικά. Πολλές ε, κυβερνήσεις κρατών μελών και η Μεγάλη Βρετανία εφάρμοσαν πολιτικές διακριτικής μεταχείρισης βάρος των πολιτών, των πολιτών τους ε, δημοσίων υπαλλήλων εξαιτία της ε, συμμετοχής τους, ε, της πολιτικής τους ιδεολογίας. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν τέτοιες πληροφορίες, οπότε υπάρχει πιθανότητα τέτοιες πληροφορίες, είπα, να διαβιβάσει τέτοιες πληροφορίες στα κράτη-μέλη σε σχέση με πολιτική τοποθέτηση πολιτών των κρατών μελών κάτι που μπορεί να διακυβεύσει την επαγγελματική σας αντιδρομία. Το αυτό συνέβη στο Λίβερ το 2009 ε, με έναν ε, υπάλληλο. Ίσως ε, θα έπρεπε να πείσουμε τα κράτη-μέλη να αποφύγουν διακρίσεις εις βάρος των πολιτών τους. Κάτι τέτοιο προϋποθέτει όμως ελευθερία του συνεταιρίζεστε. Κάτι που δεν θα ε, ε, ε, τελεσφορούσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ξέρουμε και από τη συζήτηση για τα πολιτικά κόμματα. Ο κύριος Βόξ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα καταρχάς για τον κύριο Μωράης να θυμίσω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στις ρεαλιστικές δυνατότητές μας και βέβαια αναλόγως και τις πολιτικές επιλογές που προκύπτουν. Γι' αυτό νομίζω ότι αφενός μεν πρέπει εξάπαντος να δούμε να καταγράψουμε τα πραγματικά περιστατικά για το τι είδου προγράμματα παρακολούθησε σε σχέση με τα κράτη-μέλη τρίτα κράτη μπορούν να διαπιστωθούν και να διατυπώσουμε ερωτήματα σχετικά με δεδομένα ε, συνδιαλέξεων ή επικοινωνιών και βέβαια το περιεχόμενό τους, εάν έχουν συγκεντρωθεί τέτοιου είδους στοιχεία και αναλόγως να κρίνουμε και με τις νομικές ε, βάσεις, ανάλογα με την ενόμη τι είδου ενδεχόμενη παραβίαση υπάρχει και δυνατότητα για κοινοβουλευτικό έλεγχο, προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών από τις παραβιάσεις και βασικά εκεί θα κριθεί η νομική υπόθεση εάν υπάρχει παραβίαση του δικαίου σε ποιο επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο ή σε επίπεδο χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Το γεγονός της συλλογή δεδομένων για λόγους βιομηχανικής κατασκοπίας θα πρέπει να κρυθεί κατά διαφορετικό τρόπο ασφαλώς. Και όλα αυτά τα χρειαζόμαστε προκειμένου να έχουμε μια ευκαιρία, μια δυνατότητα να διατυπώσουμε ρεαλιστικά συμπεράσματα και να δώσουμε απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών. Ευχαριστώ κυρία Ζήπεν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Το βασικό ερώτημα που μας απασχολεί και που διατυπώνουν πολύ συχνά και οι δημοσιογράφοι είναι τι είδους πόρισμα, τι είδους αποτέλεσμα μπορεί να βγει από αυτήν την Εξεταστική Επιτροπή. Οι πολιτικοί λοιπόν τις τελευταίες ημέρες ε, λένε πράγματα τα οποία με οδηγούν στο συμπέρασμα ότι πολλοί δεν θέλουν να ενημερωθούν, δεν θέλουν να μάθουν, δεν θέλουν να ρίξουν φως και κάποιοι προσπαθούν να θολώσουν τα νερά. Αν δεν τα καταφέρουν θα ήταν πράγματι πολύ ενδιαφέρον ε, γιατί με το πρίσμα παραδείγματι όταν ξέσπασε το σκάνδαλο κάποιοι είπαν «Α, ναι βέβαια χρειάζεται καλύτερη προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων ή του ιδιωτικού βίου». Ε, είναι γελίο φυσικά αν δούμε τι είδου δεδομένα και σε ποιο όγκο συλλέγονται, διαρευνώνται και συλλέγονται προσωπικά δεδομένα. Εδώ έχουμε να κάνουμε με την ε, καταπολέμηση των τρομοκρατών μας λένε και γι' αυτό δεν χρειάζεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ήδη ένας συνάδελφος σήμερα μας είπε ότι από το 2001, από τις επιθέσεις δηλαδή το Σεπτέμβριο στο World Trade Center είναι θέμα η τρομοκρατία. Ναι βεβαίως είναι θέμα η τρομοκρατία αλλά το ΕΣΕΛΟΝ προηγείται των επιθέσεων του Σεπτεμβρίου του 2001. Και έτσι είναι προφανές ότι αυτές οι παρακολουθήσεις δεν έχουν αποκλειστικό σκοπό την προστασία από, την, ε, από κάποια τρομοκρατική επίθεση, αλλά έχουν σκοπό ακόμα και τη βιομηχανική κατασκοπία. Και λυπούμε πάρα πολύ διότι δεν μπορέσαμε τελευταία εβδομάδα να συμφωνήσουμε στην άρση, στη διακοπή των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, μιας ε, εμπορικής συμφωνίας διατλαντικής και αυτό το λέω όχι γιατί δεν θέλω να συναυτεί τέτοιου είδους εμπορική συμφωνία αλλά γιατί θα πρέπει να δώσουμε λίγο χρόνο να αναλογιστούμε ποια είναι η κατάσταση διότι είναι προφανές ότι δεν μας θεωρούν φίλους οι Ηνωμένε Πολιτείες και άρα, ναι, θα, δεν θα πρέπει να σταματήσουμε να συνεργαζόμαστε με τι ΗΠΑ, αλλά θα πρέπει να δώσουμε χρόνο να αναλογιστούμε υπό ποια βάση, επί ποια βάση θα γίνεται αυτό. Και θα ήθελα πάρα πολύ σύντομα να αναφερθώ στο PNR και τη συμφωνία SWIFT με τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι αν δούμε πόσα εκατομμύρια δισεκατομμύρια προσωπικών δεδομένων καταγράφονται και συλλέγονται και δεδομένου ότι και μετά από την, ε, από την εποχή που είχαμε την Επιτροπή Έσελον έχει πολλαπλασιαστεί ο όγκος των δεδομένων, διερωτώ με, εφόσον τα στοιχεία ούτως ή άλλως τα συλλέξει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτως ή άλλως δεν έκαναν την παραμικρή προσπάθεια για ε, μία ε, θεμητή συλλογή των δεδομένων αυτών εκτός από το PNR το οποίο θα ήταν απλώς ένα ψήγμα ε, θεμητής συλλογής αφού τους άλλωστε είχαν τα στοιχεία λοιπόν γιατί να προχωρήσουμε με το PNR από ό,τι μάθαμε ε, ακόμα και επιστολές φωτογραφίζονταν όχι βέβαια το έγγραφο το ίδιο αλλά και αλλά ο φάκελος με το όνομα του αποστολέα παραλήπτη ε, φωτογραφίζονταν και αποστέλλονταν ως ψηφιακό υλικό στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών των Πολιτείων. Οπότε μπορούσε να συγκρατεί ακόμα και τα στοιχεία της ε, ταχυδρομικής επικοινωνίας. Ποιος στέλνει σε ποιον γράμμα. Λοιπόν, βεβαίως, αυτός ο μικρός κόσμος στον οποίο ζούμε, αυτό το παγκόσμιο χωριό, χρειάζεται μυστικές υπηρεσίες. Πρέπει να έχουμε μυστικές υπηρεσίες οι οποίες να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Αλλά πλέον δεν καλούνται οι μυστικές υπηρεσίες να αποτρέψουν μια ε, εμπόλεμη, μια εμπλοκή, μια σύραξη. Ε, δεν κινδυνεύουμε να βρούμε αύριο τα ρωσικά στρατεύματα πρώτων ε, πυλών. Αλλά αυτό που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες είναι να εξετάσουν στοιχεία, να αξιολογούν την χρήση των στοιχείων κτλ. Γι' αυτό λοιπόν και για να φτάσω στο τελευταίο σημείο, το ζητούμενο δεν είναι τι είδους νομοθετήματα μπορούμε να εγκρίνουμε και να επιβάλλουμε. Είναι ότι εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε την ευθύνη να διατυπώσουμε τα πολιτικά ζητήματα, να κάνουμε, να προκαλέσουμε τον δημόσιο διάλογο για την πολιτική ουσία της υπόθεσης. Και τα πολιτικά μέτρα με τα οποία μπορούμε να αποκριθούμε, να απαντήσουμε στην κατάσταση αυτή και βέβαια τις συνέπειες που μπορεί αυτά τα γεγονότα να έχουν ως προς ε, ενδεχόμενες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες που στο μέλλον μπορεί και να μην είναι καν απαραίτητε. Και εδώ αναφέρομαι όχι στην εμπορική συμφωνία για τι εμπορικέ συναλλαγέ, αλλά στη συμφωνία για το SWIFT και το PNR. Γιατί όπω είπα και νωρίτερα, δεν έχει καμιά αξία από ευρωπαϊκής πλευράς και καλό θα ήταν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να μην προχωρήσουμε σε περαιτέρω συζητήσει. Γιατί ξέρουμε ότι ε, μεταξύ μα παρακολουθούν όχι μόνο οι Ηνωμένε Πολιτείε και οι αρχέ του, αλλά και οι εθνικέ μα αρχέ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νατφέλτ. Yes, uh, Καταρχάς, θα ήθελα να επανέλθω σε κάποιες παρατηρήσεις του κύριου Κέκλοχούφου. Όντως, φαίνεται ότι σε ορισμένα σημεία συμφωνούμε. Έχουμε τελείως διαφορετική ιδέα ε, για το τι σημαίνει η δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι να ξέρουν οι πολίτες ε, τι κάνουν οι κυβερνήσεις τους. Είναι είναι έλεγχος, έλεγχος και εξουσία και έλεγχος εξουσίας. Όχι απλώς και μόνο ε, άσκηση εξουσίας από πλευράς ε, των ε, κυβερνήσεων. Διάβασα σήμερα ότι ο Πρωθυπουργό ε, του Λουξεμβούργου, ο κύριος ε, Γιούνκερ, απειλεί να παρετηθεί διότι οι κρατικές υπηρεσίες φαίνονται ότι είναι μπλεγμένε σε, σε ένα δίκτυο υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων. Εκεί φαίνεται δηλαδή ότι υπάρχει κάποια ευαισθησία, πρέπει να υπάρχει κάποια ευαισθησία και κάποια ευθύνη και το Κοινοβούλιο πρέπει να ασχοληθεί με τα θέματα αυτά. Δεν μπορούμε απλώς να βάλουμε ερωτήματα, να κάνουμε μια έρευνα ναι ή όχι. Συμφωνώ με τον Κάρλο Κουέγιο ότι θα πρέπει να στηριχθούμε και σε αυτά τα οποία έχουν γίνει ήδη μέσα στα πλαίσια της Επιτροπής Έσολων. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην διάκριση που θα κάνουμε ανάμεσα στα τέσσερα προβλήματα. Το ένα είναι η μαζική κατασκοπία εις βάρος των πολιτών, υποκλοπές και τα λοιπά, ένα σύστημα το οποίο δεν είναι ξεκάθαρο, δεν είναι σαφές και ξεπερνάει κατά πολύ την τρομοκρατία. Δεύτερον, έχουμε την κλασική κατασκοπία των ε, ΙΠΑ στις χώρες ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό είναι κάτι σαν τον James Bond. Τρίτον είναι το ότι είχαν βάλει κοριούς στα γραφεία των αντιπροσωπιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ αυτό δεν μπορώ να καταλάβω πώς συνδέεται με την τρομοκρατία, με ξεπερνάει. Ίσως είμαι αφελής, τι να σας πω. Και το τέταρτο πρόβλημα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι μαζική κατασκοπία από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών εις βάρος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρόμοια προγράμματα και συμφωνίες με τους Αμερικανούς για να ανταλλάσσονται αυτά τα στοιχεία. Δεν θέλω να θίξω ευαισθησίες, αλλά πραγματικά θα ήθελα να ξέρω ποια θα είναι, ποιες θα είναι οι συνέπειες της ε, χθεσινής δήλωσης ε, της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου ότι θα αποσυρθούν από την ε, δικαστική συνεργασία. Ε, θα πρέπει να, εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά τις συνέπειες όλων αυτών και για το PNR και για το SWIFT και για τον ασφαλή λιμένα. Ε, έγινε μια δήλωση ότι όλα αυτά θα εξεταστούν, σωστό αυτό, και ένα στοιχείο το οποίο θα πρέπει να εξετάσουμε είναι η δημοκρατική επίβλεψη των κατασκοπευτικών υπηρεσιών. Υπάρχει το INSET, το είναι ε, η ευρωπαϊκή, η παρακολούθηση αν θέλετε ε, των ε, υπηρεσιών πληροφοριών και θα πρέπει όμως να ξέρουμε. Ξέρουμε ότι δουλεύουν ε, ε, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκεί. Λοιπόν, όμως θα πρέπει να ξέρουμε ποιοι δουλεύουν εκεί, τι κάνουν ακριβώς, να υπάρχει μια δημοκρατική παρακολούθηση, αν θέλετε, μια δημοκρατική επίβλεψη των δραστηριοτήτων αυτών. Θα πρέπει να ξέρουμε τι κάνουν οι υπηρεσίες ε, πληροφοριών. Εάν έχουμε μια ευρωπαϊκή ε, υπηρεσία πληροφοριών, δηλαδή μια υπηρεσία υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καλό θα είναι, αλλά να ξέρουμε και τι κάνει. Κάποιος είπε εδώ στην αίθουσα ότι δεν θα βγάλουμε τίποτα από, την, ε, από τις μυστικές υπηρεσίες. Στην ε, Επιτροπή της CIA είχαν τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Ιταλίας. Τώρα βέβαια κάποιος είναι στη φυλακή, ο ίδιος, ο βοηθός του, δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Ε, μια πολύ σημαντική, ένα σημαντικό σημείο είναι ότι θα πρέπει να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχουμε θίξει εδώ και πάρα πολύ, πολλά χρόνια που είναι η ε, το θέμα της, ε, των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Οι Ηνωμένε Πολιτείε θεωρούν ότι η δικαιοδοσία τους απλώνεται σε, όλη την, ε, όλο τον πλανήτη. Εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο. Δεν μπορεί να ισχύει ετεροδικία, δεν μπορεί οι, οι, οι κανόνες το δίκαιο ενός ξένου κράτους, κράτους να επικρατεί, να έχει προτεραιότητα έναντι των εγχωρίων νομοθεσιών τέλος πάντων. Επίσης, γιατί να υποβάλουμε έκθεση το Δεκέμβρη και όχι τον Γενάρη, τον, τον Φεβρουάριο. Ε, γιατί να μην βάλουμε αυτούς τους δύο μήνες. Ούτως ή άλλως μέχρι το Μάρτιο έχουμε. Τελεί και μετά τελειώνει. Συμφωνώ με τις ε, παρατηρήσεις που έγιναν για τους ομιλητές. Πιστεύω ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε όσο τον περισσότερο και να υπάρχουν και κοινές συνεδριάσεις και με, εθνικούς, με εθνικά κοινοβούλια, διότι και εκεί θα γίνονται έρευνες. Ε, επί τώρα μία επίσκεψη στην Ουάσιγκτον ε, δεν βλέπω την προστιθέμενη αξία. Γιατί να πάμε στη Ουάσιγκτον, τι θα γίνει, τι θα ακούσουμε εκεί ε, που δεν θα ακούσουμε εδώ. Δεν είναι ότι έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στην διάθεσή μας. Έχω πάει πολλές φορές στη Ουάσιγκτον με μηδενικά αποτελέσματα. Γι' αυτό αυτή η επίσκεψη θα ήθελα να αφαιρεθεί από το πρόγραμμα. Ελήφθη το μήνυμα. Ο κύριο Πίρκερ. Ήρθε και η δική σα σειρά κύριε Πίρκερ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι θα πρέπει να επιδιώξουμε τουλάχιστον να καταγράψουμε τα πραγματικά περιστατικά σε σχέση με το πρίσμα και να μην συζητάμε για ισχυρισμούς μη επαληθευμένους. Να συζητούμε βέβαια ζητήματα τα οποία απασχολούν τα μέσα, αλλά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε τα πραγματικά περιστατικά πρώτα απ' όλα, δηλαδή πρέπει να διαλευκανθεί η πραγματική κατάσταση. Αλλά δεν μπορούμε να περιοριστούμε μόνο με την ανάλυση και να κάνουμε τη μία δημόσια κρόαση μετά την άλλη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διαπιστώνοντα απλώ καταστάσει. Θυμάμαι πόσε φορέ έχουμε προσκαλέσει σε δημόσια ακροάσει εμπειρογνώμονε και ε, είχαμε μόνο ένα-δύο βουλευτέ μέσα. Επομένω πρέπει και η προσέλευση από πλευρά μα να είναι ικανοποιητική. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που υπάρχει για ανάλυση της κατάστασης, αφού συγκεντρώσουμε τα πραγματικά περιστατικά, γιατί αυτό αναμένει ο κόσμος από εμά, το τι θα κάνουμε σε σχέση με τα μέτρα αυτά. Πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε αποφασιστική δράση και να εξετάσουμε, να συζητήσουμε το πώς στο μέλλον εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση θα είμαστε σε θέση να αποτρέπουμε δραστηριότητες κατασκοπίας. Μην ξεχνάμε ότι και πολιτική κατασκοπία είχαμε και βιομηχανική κατασκοπία είχαμε. Επομένως πρέπει να εξετάσουμε το πώς θα προστατευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και πώς ε, μπορούμε να προστατεύσουμε την Ευρώπη και ως χώρο βιομηχανικής παραγωγής και καινοτομίας Δεν ε, μπορούμε λοιπόν να παραγνωρίσουμε τις φωνές εκείνων των αντιευρωπαϊστών οι οποίοι ε, φωνασκούν και προσπαθούν να ε, κλείσουν το κεφάλαιο αυτό της δράσης, της αντίδρασης καλύτερα. Γι' αυτό λοιπόν ίσως θα πρέπει να συζητήσουμε ακόμα και ένα ενδεχόμενο για μια αντικατασκοπευτική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα απέτρεπε τέτοιου είδους δραστηριότητες ή θα τις προλάβαινε. Και επίσης, Ίσως θα ήταν πια η στιγμή να εξετάσουμε σε όρους τεχνικούς, τεχνολογικούς, γιατί πρέπει να περνάνε όλα τα email που στέλνουμε από τις Ηνωμένε Πολιτείε, γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα ή πώς έχουμε τη δυνατότητα να θεσπίσουμε σερβερ μεγάλους και ε, νέφος ε, ψηφιακό μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να κυκλοφορεί η πληροφορία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην περνάει από τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ε, αυτό μπορούν να μας το απαντήσουν οι ειδικοί στην τεχνολογία που θα προσκαλέσουμε ενδεχομένω. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τα πράγματα και από την εξή σκοπιά ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι εταίρο. δεν μπορούμε να του αποκόψουμε διαπαντός. Άρα λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε για το μέλλον τη δυνατότητα για μια συνεργασία ασφαλείας με κοινού κανόνε όμω. Ανάλυση, αποφασιστική και προληπτική δράση και βέβαια συνεργασία με στόχο την ασφάλεια, ενδεχομένω με μια διαφορετική μορφή και ποιότητα για το μέλλον. Αυτή θα ήταν η πρότασή μου συμπληρωματικά στα όσα υπόθηκαν ήδη Πάντω ε, πάντως θα ήθελα να ε, ε, κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Θα ήταν μεγάλο λάθος να ασχοληθούμε μόνο με την ανάλυση και να μην διατυπώσουμε τα συμπεράσματα. Θα πρέπει να, είμαστε θέση να διατυπώσουμε συγκεκριμένα και επικοδομητικά ε, συμπεράσματα για το μέλλον. Για το πώς μπορεί η Ευρώπη να προστατευθεί από την υποκλοπή και μεταφορά δεδομένων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενο ομιλητή. Πρόεδρε, νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη για τεχεία δράση και μελέτη της κατάστασης των δυνατών πιο γρήγορα. Αυτή τη στιγμή έχουμε εφημερίδες που με άρθρα ή φήμες που κυκλοφορούν δείχνουν ίσως μόνο την κορφή του παγόβουνου, αλλά στοιχεία δεν έχουμε. Και είναι πολύ σημαντικό να συλλέξουμε τα στοιχεία και τα ντοκουμέντα αυτά που χρειάζονται. Ως εκ τούτου λοιπόν ε, η Επιτροπή Διατλαντικής Συνεργασίας και η κυρία Μάλστρομ έχουν πολύ μεγάλη σημασία αλλά μεγάλο, ε, το, το πιο σημαντικό θα είναι η δική μας εξεταστική επιτροπή να είναι σε θέση να ε, διερευνήσει την κατάσταση έτσι ώστε να αποκαταστήσει τα πραγματικά παραστατικά, να μπορεί να δει την πραγματική τη ροή των γεγονότων. Επίσης πολύ σημαντικό είναι πριν τις ε, διακοπές να μας χορηγηθεί ένα υπόμνημα με μια συνοπτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων της Επιτροπής Έσλων για να δούμε σε τι αποτελέσματα έχει καταλήξει και να συνεχίσουμε ουσιαστικά το έργο αυτό. Να αξιοποιήσουμε μη τι άλλο το έργο που έχει γίνει. Επίσης και λόγω των θερινών διακοπών επήγει πολύ να αναπτύξουμε, να αναλάβουμε τις επαφές με τα εθνικά κοινοβούλια και θα προτιμούσα πριν να κλείσουμε για το καλοκαίρι ε, να έχουμε ήδη κάνει μια πρώτη επαφή για να ζητήσουμε τη συνεργασία. Αλλά πρέπει να πούμε επίση ότι εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με μυστικέ υπηρεσίε. Έχουμε να κάνουμε πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε να κάνουμε με συσχετισμό τη στρατιωτική με την βιομηχανική διάσταση και σε αυτό πρέπει να πω ότι δεν έχουμε αρκετά στοιχεία. Ε, γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να προσκαλέσουμε και εμπειρογνώμονε οι οποίοι είναι σε θέση να ε, διαβάσουν αυτού του συσχετισμού ε, από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα ενδεχομένως που έχουν την πρωτοπορία στον χώρο αυτόν για να δούμε η οικονομική με την στρατιωτική διάσταση πώς αναμειγνύονται και τι είδους ε, συνέπειες μπορεί να έχουν αυτά και για τις ελευθερίες και για την ε, οικονομία μας. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η διάσταση, δεν μπορούμε να την υποβιβάσουμε και παρακαλώ να συμπεριληφθεί και αυτή στο πεδίο εξέτασης. Και επίσης κύριε Πρόεδρε θα ήταν χρήσιμο να, να έχουμε επαφές και με ιδιωτικές επιχειρήσεις που έχουν δραστηριοποιηθεί στο τομέα αυτών. Επίσης μιλούμε για συνεργασία με εθνικά κοινοβούλια μέσα στην Ευρω... της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά νομίζω θα ήταν χρήσιμο να συναντηθούμε και με συναδέλφους από το ΗΠΑ, από το Κογκρέσο, γιατί ασφαλώς θα υπάρχουν κάποιοι οποίοι ε, μεριμνούν για την προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών, των πολιτικών ελευθεριών, που είχαν αντιδράσει στο πρίσμα. Ε, άρα λοιπόν πρέπει να στραφούμε προς αυτούς τους συναδέλφους μας στην άλλη όχθη του Ατλαντικού. Σας ευχαριστώ κυρία Λάτφορτ. Ευχαριστώ. Επανέρχομαι στις παρατηρήσεις του κυρίου Κόελλο. Έριξα μια ματιά στην έκθεση της Επιτροπής Εσελών όσο συζητούσαμε και πραγματικά έχω την αίσθηση ότι το έχουμε ξαναδεί αυτό το θέμα. Διαβάζοντας τα πορίσματα και τις συστάσεις της Επιτροπής Εσελών και πραγματικά ε, πολύ σωστές ήταν οι παρατηρήσεις του Κάρλος ότι οι συστάσεις της Επιτροπής σελών δεν ε, εφαρμόστηκαν. Και είναι πολύ εύστοχες παρόλα αυτά και οι συστάσει και τα πορίσματα της Επιτροπής Εσελών. Δεν θέλω να με παρεξηγήσετε. Ελπίζω ότι η... η συγκέντρωση των πραγματικών περιστατικών και χαρτογράφηση θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατόν. Γιατί φοβάμαι ότι πολύ γρήγορα θα φτάσουμε το Μάιο ή ακόμη και νωρίτερα τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο να μην έχουμε ε, φτάσει στην ε, ουσία του πράγματος, δηλαδή στην άντληση των πολιτικών και νομικών ε, συμπερασμάτων. Βέβαια, τους τελευταίους μήνες, για να μην πω και χρόνια, πολλά έχουν υποθεί και γραφτεί για όλα αυτά και σίγουρα έχουμε πολλά ακόμη να μελετήσουμε, αλλά ήδη έχουμε κάποιες αδερές γραμμές ό,τι αφορά αυτά τα, τα ζητήματα της μαζικής παρακολούθησης στην αρχή έγινε με βάση την αρχή ε, μόνο αλλοδαπούς αφορά και δεν ενδιαφέρει τους ε, νομοθέτες μας. Αλλά κάτι τέτοιο είχε υποθεί και στην Επιτροπή και στην έκθεση Επιτροπής Σελών. Είχε επισημαθεί και αυτό το θέμα. Θα πρέπει ε, να δούμε τι γίνεται και με τα Εθνικά Κοινοβούλια εφόσον έχουν επιτροπές εποπτείας για θέματα αυτά. Και η Επιτροπή του Westminster επιτέλους έχει συσταθεί και ε, μιλά, ε, δεν θα πρέπει να είναι κανείς ε, κριτής και κρινόμενος. γιατί στην αρχή ήταν μέλη της εκτελεστικής εξουσίας που συμμετείχα στην εποπτεία αυτή. Δεν είναι σωστό αυτό. Και όπως είπα στην, και την περασμένη εβδομάδα, περιμένω με κομμένη την ανάσα την, τα πορίσματα της Επιτροπής Έρευνας του Westminster για την διαλεύκανση των δραστηριοτήτων των μυστικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν θεωρώ ότι θα τα μάθουμε όλα, αλλά να μην αναλωθούμε σε πολύμηνη συγκέντρωση πληροφοριών και σε πολλές λεπτομέρειες και χάνοντας, επιμένοντας τα δέντρα χάσουμε το δάσος. Επίσης, και σε ό,τι αφορά τις διαπραγματεύσεις για την ανταλλαγή των δεδομένων, πώς θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσει για το πακέτο αυτό. Είναι σημαντικό να το λάβουμε υπόψη για την νομοθεσία που θα καταρτήσουμε και τις διπλωματικές και πολιτικές σχέσεις που θα έχουμε με τους εταίρους μας. Καλή τύχη εύχομαι στον ε, εισηγητή της έκθεσης, γιατί πραγματικά θα είναι κολοσιαίο το εγχείρημα αλλά θα πρέπει το συντομότερο δυνατόν να περάσουμε χωρίς να δηλήσουμε τον κόνοπα, γιατί δεν πρόκειται να αναλύσουμε και την παραμικρή λεπτομέρεια. Ήδη τις βασικές γραμμές τις γνωρίζουμε. Θα πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια συμπεράσματα για να μην έχει και η έκθεση αυτή τη δίχη που είχε η έκθεση της Επιτροπής Σελών. Ναι, είναι, είναι προφανές ότι πολλές παρατηρήσεις ε, αφορούν το χρονοδιάγραμμα. Συνειδητοποιούμε ότι το θέμα μας είναι τεράστιο, που δεν μπορεί να εξαντληθεί μέχρι το τέλος της θητείας. Αλλά επιμένω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και αυτό το θέμα έχει ε, κινητοποιήσει όλους τους πολίτες. Ε, ε, οι πολίτες περιμένουν κάτι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να τους προσφέρουμε μια σημαντική και μια ουσιαστική απάντηση μέχρι το τέλος της θητείας μας. Γι' αυτό ακριβώς είχαμε θέσει και το χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του χρόνου έτσι ώστε στις αρχές του 2014 να είμαστε στην τελική ευθεία. Γιατί ούτως ή άλλως ε, είναι και η προεκλογική εκστρατεία το 2014. Βέβαια, μπορούμε να μην ολοκληρώσουμε μέχρι το τέλος του 2013 και θα το δούμε και στην διάσκεψη των Προέδρων. Όμως ας κάνουμε ό,τι μπορούμε, ας καταβάλουμε καθόλου την προσπάθεια τους επόμενους μήνες να εργαστούμε ε, εντατικά, να έχουμε μια στρατηγική, να καταστρώσουμε μια στρατηγική έτσι ώστε το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να ε, εποφεληθούμε στο δυνατόν περισσότερο από το χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορούμε να ε, εποφεληθούμε και από τις ολομέλειες του Στρασβούργου. Ε, ας δούμε και ποιες είναι και οι πληροφορίες που έχουν μαζέψει τα κράτη-μέλη και θα δούμε τι θα γίνει. Κύριε Σταβάρες, ευχαριστώ Πρόεδρε. Εμείς ενώνουμε τώρα τα κομμάτια του παζλ και αυτό δεν είναι και δύσκολο βέβαια γιατί τα κομμάτια του παζλ ταιριάζουν μεταξύ τους. Το PNR, το SWIFT, Echelon και τώρα το Prisma. Ε, θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι όταν ασχολούμεθα με το PNR και το SWIFT οι Αμερικανικές αρχές έλεγαν ότι εμείς ε, δεν θα εκμεταλλευτούμε τις πληροφορίες αυτές. Τώρα όμως βλέπουμε το Prisma και ε, μας λένε ότι δεν ακούμε κάθε τηλεφωνική συνδιάλεξη ξεχωριστά. Ε, απλώς το pattern θέλουμε να ε, δημιουργήσουμε. Επομένως, βλέπουμε ότι όλα αυτά ταιριάζουν ε, και η λογική τους είναι κοινή και συνδυάζονται μαζί τους. Δεν χρειάζεται να εκμεταλλεύονται να βλέπουν τις, ε, τα δεδομένα από ένα, από μία ενέργεια, ε, απλώς τις συλλέγουν και τις εκμεταλλεύονται με το άλλο σύστημα. Τέλος πάντων, το πρόβλημα είναι ότι οι δηλώσεις που κάνουν οι κυβερνήσεις, είτε είναι δικές μας είτε είναι ξένες, δεν είναι ειλικρινείς, είναι υποκριτές. Είδατε τι έγινε με το αεροπλάνο την προηγούμενη εβδομάδα. Ο υπουργό μας μας είπε ότι είχε τεχνικό πρόβλημα το αεροπλάνο του Εύω Μοράλες και γι' αυτό δεν μπορούσε να προσγειωθήσει στην Πορτογαλία. Λοιπόν, όταν, όταν όμως είχαμε τις απαγωγές ε, των ε, υπόπτων από πλευράς Αμερικανών, κανένα αεροπλάνο δεν είχε ε, τεχνικό πρόβλημα. Τώρα ο πρόεδρος ε, της ε, Βολιβία, ε, που το προεδρικό αεροπλάνο του προέδρου της Βολιβία που ήθελε να περάσει από την Πορτογαλία είχε τεχνικό πρόβλημα. Τέλος πάντων, πρέπει να είμαστε ειλικρινεί, να μην, να μην δεχόμαστε αυτέ τι υποκρισίες και να μην, σκανδαλιζό, να μην σκανδαλιζόμαστε από αυτά τα οποία λένε. Υπάρχει, όπως είπε και ο κύριος Κουέλιο, ε, έχουμε ένα ψήφισμα όσον αφορά τις ε, ρήτρε διασφάλισης ε, που αφορούν την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην ανταλλαγή πληροφοριών. Και η απάντηση της Αντιπροέδρου Ρέντινγκ ήταν ότι η απάντηση εδώ στην Ολομέλεια και δεν πρόκειται να δοθεί συνέχεια. Τώρα υπάρχει ένα ψήφισμα για το πρίσμο λέμε στο σημείο 15 ε, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή αντιστοιχία όσον αφορά τις μικτές επιτροπές ε, νομικής, νομικές και ε, δικαστικές όσον αφορά την προστασία των δεδομένων. Εμείς δεν έχουμε τρόπο να ελέγχουμε την, ε, τις προφορίες ε, που μας δίνει η Europol. Με τη Europol όμως τι γίνεται. Εάν η Europol δίνει πληροφορίες εμάς ή στην κυρία Ρέντινγκ, όπου υποθέτω ότι κάνει, το κάνει. Δεν ξέρουμε αν ο Σνόουντεν είναι ήρωας ή προδότης, αλλά το, οι πολίτες πρέπει να παίρνουν, αυτές, αυτή, να τις αποφάσεις. Γι' αυτό είμαστε και εμείς εδώ. Και έγινε μια αλλαγή στις έρευνες. Εμείς δεν θα πρέπει να ε, παίξουμε την ίδια χορογραφία όπως στο παρελθόν, όπου υποπτευόμαστε κάτι, μετά ανακαλύπτουμε την αλήθεια, μετά κάνουμε ένα σκάνδαλο, μετά ερευνούμε, ερευνούμε και μετά δεχόμαστε να συνεχίσουμε όλες αυτές τις δραστηριότητες, να μην συνέβαινε τίποτα. Και το κάνουμε και εμείς μετά. Και μετά το αμερικανικό SWIFT υπάρχει ένα ευρωπαϊκό SWIFT και μετά το αμερικανικό PNR έχουμε και ένα ευρωπαϊκό PNR. Λοιπόν, επομένως τι χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε έρευνα, μου αρέσουν οι έρευνες, όμως μετά πρέπει να υπάρχουν και κάποιες πολιτικές συνέπειες, γιατί με αυτόν τον τρόπο μόνο θα μπορέσουμε να, να ακουστούμε. Γι' αυτό θα πρέπει το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο να ε, ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Ευχαριστώ κύριε Ρομέρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να επιμείνω στην κοινοβουλευτική διάσταση αυτής της ερευνητικής επιτροπής. Γιατί σε τελική ανάλυση αυτό που περιμένουν οι συμπολίτες μας και ψηφοφόροι μας από εμά είναι να διαλευκάνουμε τη, τα γεγονότα, τα περιστατικά αυτά. Και με τους προσκεκλημένους σε αυτή την εξεταστική επιτροπή, εκπροσώπους μυστικών υπηρεσιών ή επίσημων οργανώσεων, οι πληροφορίες από αυτούς τους ανθρώπους θα, θα είναι ελάχιστες. Θα πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε ε, την παρουσία των ε, Αμερικανών γερουσιαστών. Γιατί δεν έχουν όλοι, όλα τα μέλη του Κογκρέσου την ίδια γνώμη στις Ηνωμένε Πολιτείε. Συμφωνώ με την κυρία Ίντβελτ για την αποστολή μας στη Ουάσιγκτον. Έχουμε α, ε, ταξιδεύσει πολλές φορές για το SWIFT, για το PNR, για όλες τις πολιτικές προστασίες των δεδομένων. Και είχαμε πάντα συναντήσεις με την κυβέρνηση, με εκπροσώπους της κυβέρνησης και όχι με, τους, με τα μέλη του Κογκρέσου. Ενώ όταν είχαμε επαφές εδώ με τα μέλη του Κογκρέσου μας είπαν ότι ε, απαγορεύεται σε αυτούς να ταξιδέψουν στην Αλλοδαπή γιατί δεσμεύονται από το απόρριτο και μάλιστα υπάρχει και στο Κογκρέσο μία επιτροπή ε, για επίσημα μυστικά ή επίσημα απόρριτα, κάτι που δεν έχουμε εμείς. Οπότε δεν ξέρουμε από, από το Αμερικανικό Κογκρέσο ποια ήταν η αντίδραση, όχι τώρα, αλλά στο παρελθόν. Όπως μας είπε πολύ σωστά ο κύριος Κοέγιο, δεν είναι κάτι καινούριο και πρωτοφανέ. Και αυτή η ανακάλυψη της παγκοσμιοποίησης, της μαζικής παρακολούθησης και του δυσανάλογου χαρακτήρα μας έχει προβληματίσει κάπως και από προσανατολίσει Αλλά δεν είναι καινούριο αυτό το φαινόμενο. Να ενισχύσουμε λοιπόν την κοινοβουλευτική διάσταση και να εξετάσουμε αυτά τα θέματα με τα μέρη του Κογκρέσου για να δούμε γιατί φτάσαμε εδώ. Ξέρουμε ε, την προέλευση των νομοθεσιών των ΗΠΑ και ξέρουμε και τη στρατηγική τους και ε, εκείνοι δεν γνωρίζουν ε, πάντα τις δικές μας νομοθεσίες ή τις δικές μας ε, αντιλήψεις περί ιδιωτικής σφαίρας. Υπάρχει ένα έλλειμμα διαλόγου εδώ και φτάσαμε σε ένα δύσκολο σημείο. Γιατί θα πρέπει εμείς ως ευρωβουλευτές ε, να συγκεντρώσουμε πληροφορίες από ανθρώπους που δεν έχουν διασυνδέσεις με τις κυβερνήσεις. Κύριε έφυγε ο Κύρκοπ δεν ε, έχουν πεθάνει οι πληροφοριοδότες που μας πρότεινε ο κύριος ε, Άλμπρεκτ, γιατί μας ενδιαφέρουν αυτά τα στοιχεία. Και μπορούμε να συγκεντρώσουμε και τέτοιες πληροφορίε. Αλλά όταν προετοιμάσαμε το πακέτο με την οδηγία και τον κανονισμό, είχαν έρθει εδώ και μας ενημέρωσαν πρώην εργαζόμενοι στην Google, στη Microsoft. Γιατί τέτοιε πληροφορίε θα πρέπει να συγκεντρώσουμε. Και τέτοιες πληροφορίες θα μας τις, δώσουν ακαδημαϊκοί, πανεπιστημιακοί, εμπειρογνώμονες, πληροφοριοδότες φυσικά, επιχειρήσεις, γιατί μόνο από εκπροσώπους των κυβερνήσεων οι πληροφορίες που θα λάβουμε θα είναι αδιαφανείς. Είναι δεδομένο από τη φύση των μυστικών υπηρεσιών. Και σίγουρα με τέτοιες μονοπληροφορίες δεν πρόκειται να σημειώσουμε πρόοδο φως θα χυθεί μόνο από πληροφορίες των βουλευτών, από πληροφοριοδότες, από πανεπιστημιακούς. Οπότε μερικές φορές είχαμε και συναντήσει με εθνικά κοινοβούλια, αλλά και στις συνελεύσεις αυτές ελάχιστη η πρόοδος σημειώθηκε. Αν γνωρίζουμε όμως ότι υπάρχουν εθνικοί βουλευτές που είναι εμπειρογνώμονες και ασχολούνται με τα θέματα αυτά, τότε θα ήταν ενδιαφέρον να τους καλέσουμε στην Ερευνητική Επιτροπή για να μας ενημερώσουν. Γιατί ίσως υπάρχουν και παράλληλες επιτροπές στα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Στη Γερμανική Βουλή, στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, στα κοινοβούλια των χωρών ε, της Μεγάλης Βρετανίας υπάρχουν εμπειρογνώμονες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Γιατί θα ήταν σημαντικό σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να έχουμε σχέση μαζί τους. Και υπάρχει διαφορά στις αντιλήψεις, γιατί ε, για ορισμένους ε, ε, είναι η παροχή πληροφοριών προδοσία, για μας είναι απλώς καταγγελία. Το θέμα του whistleblower, του πληροφοριοδότη, είναι αγγλοσαξονική κουλτούρα. Γιατί για ε, καταγγελίες ε, φορολογικών παραδείσων και φοροδιαφυγής είναι καλές οι καταγγελίες και ο πληροφοριοδότης ε, κάνει ευάρεστο έργο. Αν μας καταγγέλει παράνομη δραστηριότητα μυστικών υπηρεσιών τότε γίνεται προδότης. Θα πρέπει να δώσουμε μια απάντηση. Δεν είμαστε εμείς οι κυβερνήσεις, εμείς είμαστε ευρωβουλευτές. Θα πρέπει να πούμε στους Ευρωπαίους πολίτες ότι αν χαράξουμε αντιτρομοκρατική στρατηγική, οφείλουμε να του ενημερώσουμε και να ξέρουν τι είναι. Και αν είναι άλοθη αυτό η αντιτρομοκρατική στρατηγική, και αυτό δικαιούνται να το μάθουν οι πολίτε. Σε αυτό το συμπέρασμα θα πρέπει να καταλήξουμε όταν ολοκληρώσουμε την έκθεση που δεν θα είναι σίγουρα οριστική, αλλά σίγουρα θα μας φέρει πιο κοντά σε μια στρατηγική που θα πρέπει να είναι σοβαρή και να έχουμε ένα γνήσιο διάλογο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Δια μέρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε τι εντολή μας έχει δώσει το ψήφισμα της Ολομέλειας. Η εντολή είναι σαφέστατη. Περιορίζεται σε πέντε θέματα. Έρευνα, πρώτον. Δεύτερον, εντοπισμός των ευθυνών. Τρίτον, συνέπειες της υποτιθέμενη κατασκοπίας ή παρακολούθησης στην ιδιωτική σφαίρα και την, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τέταρτον, νομικό θέμα των ένδικων μέσων, των προσφυγών και των αποζημιώσεων, ανάλυση ζημιών και κινδύνων και τέλος συστάσεις. Πώς θα τα κάνουμε όλα αυτά. Είναι σαφώς οριοθετημένη η εντολή της Ολομέλειας προς την Επιτροπή. Θα ήθελα να πω στην κυρία Λάτφορτ ότι συμφωνώ ότι το εφικτό είναι ο εχθρός του καλύτερου. Πολλό δε μάλλον που έχουμε πολύ στενό χρονικό ορίζοντα. Έχουμε πολύ περιορισμένο χρονοδιάγραμμα για να ολοκληρώσουμε όλες αυτές τις αποστολές και τα καθήκοντα. Εγώ θα προτιμούσα το εξής. Να προσδιορίσουμε τους καλεσμένους και τις ακροάσεις και να μην ε, ε, θέλουμε να είμαστε υπερβολικά σχολαστικοί και εξαντλητικοί. Εγώ θα προτιμούσα πρώτα να καλέσουμε τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, πρώτο και τελευταίο. Δηλαδή, να έρθει στην αρχή των εργασιών της Επιτροπής και στο τέλος των εργασιών της Ερευνητικής Επιτροπής. Αυτό θα έχει ένα πολύ σημαντικό πολιτικό αποτέλεσμα και αντίκτυπο. Γιατί αυτό που θέλουμε να πούμε στους πολίτες που τους αναφέρουμε συχνά είναι προειδοποίηση, πρώτον. Δεύτερον, πολιτική διαμαρτυρία. Τρίτον, ε, να επιστήσουμε την προσοχή. Και τέταρτον, να απαιτήσουμε απόδοση ευθυνών. Εγώ έχω κάποια πείρα στα πλαίσια των εξεταστικών επιτροπών. Έχω την αίσθηση ότι το χειρότερο που θα μπορούσε να μας συμβεί και ο μεγαλύτερος εχθρός της αποτελεσματικότητας είναι η υπερβολική σχολαστικότητα και η φιλοδοξία να είμαστε εξαντλητικοί. Αυτό να το προσέξουμε στους καλεσμένους, στις ακροάσεις, στα χρονοδιαγράμματα και φυσικά να ορίσουμε από τώρα πότε θα πρέπει να καταλήξουμε σε συστάσεις. Κύριε Δρούσα, έχετε το λόγο. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι λίγο μπλεγμένος ακούγοντας όλων των, όλους τους Ο καθένας έχει τις απόψεις του βέβαια. Εγώ δεν θα είμαι πολύ θετικός ε, στις, ε, στην παρέμβασή μου και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων διότι ίσως ε, φανήσα να κριτική. Ξεκινώντας με μια πρώτη παρατήρηση είναι ότι νομίζω ότι έχουμε χάσει το δυναμισμό μας και αυτό μην το υποτιμάμε. Να σας πω πώς αισθάνθηκα τις τελευταίες μέρες, κυρίως όταν ασχοληθήκαμε με το θέμα αυτό στο Στρασβούργο. Έχει να κάνει και όλες και με την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Και μην ανησυχείτε, δεν θέλω να ανοίξω τη συζήτηση προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά να σας πω πώς αισθάνθηκα. Συζητάγαμε στην Ολομέλεια ένα ψήφισμα σαν αντίδραση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα όσα συνέβησαν, σε όσα ακούσαμε από τα άρθρα στον τύπο. Είπατε ότι η ευρωπαϊκή κοινή γνώμη είχε σοκαριστεί και όλα αυτά. Και τι έγινε την μέρα πριν να ψηφίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το δικό του ψήφισμα, ήδη υπήρχαν δηλώσεις από ηγέτες κάποιων κρατών μελών ή από, ενός, από ένα κράτος μέλος που μετά, και μετά είχαμε ε, και δήλωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις ε, για την συμφωνία ε, για την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είπα, χωρίς καν να περιμένουν ε, το τι θα πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν θέλω να υπερτιμήσω το ρόλο μας, αλλά πραγματικά θέλω να σας πω πώς αισθάνθηκα. Δηλαδή, από τη μια είχαμε ένα χαστούκι με τα όσα συνέβησαν από τις Ηνωμένε Πολιτείες, από όσα έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείες και μετά όμως έφαγε κι άλλο ένα χαστούκι από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, τα οποία δεν σεβάστηκαν αυτό το οποίο έπρεπε να κάνουμε εμείς και δεν περίμεναν να δουν τι θα κάνουμε. Τα λέω όλα αυτά γιατί πρέπει να ε, βάλουμε μια κάποια ισορροπία αν θέλετε σε αυτά τα οποία θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε και, και θα κάνουμε στο τέλος. Επίσης κάποια ερωτηματικά σαν βάση και των συζητήσεων που είχαμε μέχρι τώρα. Καταρχάς ποιος είναι ο στόχος αυτής της έρευνας τα κάνουμε αυτά για τα μέσα μαζικής ε, ενημέρωσης για να φανεί ότι αντιδρούμε ή το κάνουμε για την ουσία. Ελπίζω ότι το κάνουμε και να συμφωνούμε όλοι, το κάνουμε για την ουσία. Φοβάμαι όμως ότι δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες. Η Κάρμεν Ρομέρο το είπε πάρα πολύ εύγλωτα, αλλά και άλλοι ανέφεραν στο γεγονός ότι οι πολίτες ε, πρέπει να ενημερωθούν, έχουν δικαίωμα στην ενημέρωση. Οι κυβερνήσεις δεν το κάνουν, αλλά θα το κάνουμε εμείς. Αλλά αν το κάνουμε όμως, πρέπει να το κάνουμε σωστά, έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε κάποιες προσδοκίες, τις οποίες μετά δεν, μπορέσουμε, δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε. Και η ζημιά για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για το στάτους του, για το γόητρό του, για την θέση του, για την αξιοπρέπειά του, θα είναι μεγάλη. Είπαμε επίσης ότι χρειαζόμαστε αποτελέσματα και μετά πρέπει να δούμε και τις συνέπειες. Και διαρωτώ αυτές οι συνέπειες ποιες θα είναι, τι αρμοδιότητες έχουμε έτσι ώστε να μπορούμε να μιλάμε για τις ε, συνέπειες. Επομένως, τι θέλω να πω, ότι θα πρέπει από την αρχή να θέσουμε έναν σαφή στόχο Ποιος είναι ο σκοπός μας, τι θέλουμε να πετύχουμε σαν αποτέλεσμα αυτής της έρευνας. Και μετά θα πρέπει να κοινοποιήσουμε, να ανακοινώσουμε το στόχο αυτό με τον σωστό τρόπο έτσι ώστε να μην δημιουργήσουμε προσδοκίες τις οποίες δεν θα μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε. Τώρα όσον αφορά τις αρμοδιότητες θα ήθελα να έχουμε μία παρουσίαση που θα παρουσιάζει τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στον τομέα αυτό. Έχουμε αρμοδιότητες. Έχουμε καμία αρμοδιότητα να το κάνουμε, έτσι ώστε να δούμε και ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα ή η συνέπεια. Μετά, η ικανότητά μας. Μπορούμε να το κάνουμε. Ακούσαμε πολλά σχετικά με το πρόγραμμα εργασίας. Και διαρωτώ με κάθε σεβασμό, μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Ξέρουμε ότι έχουμε πάρα πολύ δουλειά και μετά άλλα σημεία. Επομένως, συμφωνώ με αυτά που είπε η Κορνίλια, θα πρέπει ίσως να σκεφτούμε, να δημιουργήσουμε μια παράλληλη δομή αν χρειάζεται. Ένας άλλος συνάδελφος εξέφρασε ένα φόβο με τον οποίο συμφωνώ. Δηλαδή ότι υπάρχει ο κίνδυνος αυτός, υπάρχει ο κίνδυνος ότι όλο αυτό το θέμα θα φιλορροήσει και δεν θα πηγαίνει κανείς στην ομάδα στο τέλος. Και ε, επομένως και εκεί η αξιοπιστία μας και η αξιοπρέπειά μας ε, ε, βρίσκεται σε κίνδυνο. Και εν κατακλείδη πρόεδρε, οι προσκλήσεις... Ακούστηκε να καλέσουμε τον Αμερικανό πρέσβη. Αυτό είναι. Αυτό είναι από αμερικανικής πλευράς να έρθει μόνο πρέσβης και να μας πει τι. Ήδη όλοι ξέρουμε τι θα μας πει. Να σας τα πω κι εγώ. Είτε έρθει στο τέλος, είτε έρθει στην αρχή, απόλυτα δίκαιο έχετε, αλλά αυτός θα είναι ο στόχος της Επιτροπής. Να έχουμε τον Αμερικάνο πρεσβευτή εδώ. Η πρόταση να συμπεριληφθούν μέλη του Κογκρέσου είναι πάρα πολύ σημαντική. Επίσης θα έκανα και ένα βήμα ακόμα. Αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών και από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και ε, από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και, Πρόεδρε, όσον αφορά τις προσκλήσεις. Ίσως να είναι προκλητικό, να ακουστεί προκλητικό. Αλλά άκουσα ε, στο Στρασβούργο μια συνάδελφο να λέει γιατί να μην και τον πρόεδρο Ομπάμα άκουσα κάποιες αντιδράσεις ότι είσαι τρελή, είσαι τι λες. Ναι, ίσως είναι τρελή ιδέα, δεν λέω, αλλά είναι ένα σημείο αυτό ότι με τον τρόπο αυτό κάνεις μια δήλωση, κάνεις ένα statement. Δεν πρέπει να να, να, να, να, να διστάσουμε, δεν θα πρέπει να διστάσουμε να καλέσουμε και ανθρώπους που μπορεί και να μην έρθουν, αλλά και το ότι δεν θα έρθουν θα σημαίνει κάτι θα είναι ένα μήνυμα το οποίο θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε. Και με τον κύριο Σνόουντεν κτλ. κτλ. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τελευταία παρατήρηση. Εξωτερική πολιτική. Ξέρω ότι δεν είναι της Επιτροπής μας αυτό το θέμα, αλλά και όταν μιλάμε για στόχο και για τα αποτελέσματα και για τις συνέπειες, θα πρέπει να έχουμε και μία πλήρη συζήτηση όλα αυτά τι θα σημαίνουν για την εξωτερική πολιτική μας και για τις σχέσεις ε, με, την Ευρωπαϊ... με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και απέναντι στην αξιοπιστία και μελλοντική αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος άνευ μικροφώνου. Κύριος Βότσαν και μετά κύριος Μπουργκέτσιο, αλλά θα ήθελα να σας ε, καθιστάσω ότι όντως πιστεύω πως δεν πρόκειται να αφήσουμε να ξεφουσκώσει όλο αυτό το μεγάλο θέμα. Ίσως να μπορέσουμε να το εξαντλήσουμε, αλλά έχουμε και ένα τεράστιο καθήκον, πολιτικό, κοινοβουλευτικό. Και πρέπει ως εκ τούτου να αξιολογήσουμε όχι μόνο τις συνέπειες όλης αυτής της υπόθεσης των αποκαλύψεων για το πρίσμα, τις ευθύνες ε, και πάνω απ' όλα την αξιοπιστία της ε, αμερικανικής κυβέρνησης των Αμερικανικών αρχών ως εταίρων αξιόπιστων. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι είχαμε και σοβαρές, σοβαρά θέματα που διαπραγματευόμαστε, παραδείγματι ε, μια συμφωνία για τις επενδύσεις και το, τις εμπορικές συναλλαγές, αλλά και τα δικαιώματα των πολιτών. Και πρέπει και από κοινοβουλευτική άποψη να τα αξιολογήσουμε. Πρέπει να αξιολογήσουμε δηλαδή όλα αυτά τα μαζικά προγράμματα κατασκοπίας παρακολούθησης εις βάρον Ευρωπαίων πολιτών, σε ποιο βαθμό πράγματι ε, είχαν να κάνουν την προστασία από την τρομοκρατία, μια εσωτερική ε, στρατηγική προστασία ή καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Γιατί, γιατί από αυτές τις μαζικές πρακτικές επιτήρησης, ε, παρακολούθησης πολιτών, δεν μπορούμε φυσικά να ε, αγνοήσουμε την ανάγκη για την προστασία από την τρομοκρατία. Αυτό είναι το καθήκον μας ως βουλευτών και πρέπει βεβαίως να δώσουμε περιθώριο για συζήτηση, για παρουσίαση και έκθεση της κατάστασης και στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Και προτείνω, επιμένω, αυτές οι επαφές να ξεκινήσουν αμέσως από το Σεπτέμβριο και δύο από τις 5 του μηνός. Ο κύριος Βότσον έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Εγώ ξέρω ότι έχω στην εκλογική μου περιφέρεια, ε, το, στο Τσέλτναμ συγκεκριμένα, τα ε, κεντρικά γραφεία της υπηρεσίας αντικατασκοπίας, αλλά και το τεμπούρα στο μπουτ της Κορνουάλης, που έχει να κάνει με τι επαφέ με τι ΗΠΑ και ξέρετε ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής αυτής πριν από 12 χρόνια όταν ξεκίνησε η έρευνα για το Echelon είχα ασχοληθεί πολύ ενεργά με το θέμα αυτό. Κύριε Πρόεδρε, η συλλογή δεδομένων είναι το πρώτο κεφάλαιο στο βασικό εγχειρίδιο λειτουργία κάθε ε, αντικατασκοπευτική υπηρεσία κάθε καθεμιστικές υπηρεσίες. Το θέμα είναι τώρα πια έχουμε προχωρήσει περισσότερο ως προς τις νομικές έννοιες. Και μετά το άρθρο 12 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ανθρώπινων Δικαιώματα που λέει ότι δεν μπορεί κανείς να υπάγεται σε ε, αυθαίρετη παρέμβαση στον οικογενειακό του βίο, τον ιδιωτικό του βίο, τον οίκο του ή την αλληλογραφία του και αυτό βεβαίω στο άρθρο 8 στη Σύμβαση, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα όπου αναφέρεται ότι δεν μπορεί να υπάρχει παρέμβαση ως προς την ιδιωτικότητα της, ε, των επικοινωνιών παρά μόνο για λόγους που ορίζει ο νόμος και προστασίας ε, της εθνικής ασφάλειας και παραπέρα με το χάρτη των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων που αναπτύσσεται περισσότερο το θέμα λέμε ότι αν υπάρξει ανάγκη για επεξεργασία δεδομένων θα πρέπει με τρόπο ε, θεμητό και επί τη βάση που ορίζει ο νόμος να γίνεται αυτή. Η συλλογή λοιπόν δεδομένων, Πρόεδρε, με τον τρόπο που ε, διεξάγεται είναι προς το συμφέρον του, της δημοσίας ασφάλειας και ε, με, ο, τρόπος με τον οποίο ε, λειτουργούν ε, οι τρομοκράτες, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει πολύ προωθημένη τεχνολογία, ασφαλώς χρειάζεται μια αντίστοιχη ανταπόκριση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι θεμητή η παρέμβαση των κρατικών υπηρεσιών. Θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο έχουν παρακολουθήσει οι εθνικές αρχές τους ε, υπηκόους άλλων κρατών, αλλά ταυτόχρονα και σε ποιο βαθμό έχουν ξεπεράσει αυτές οι αρχές τη βασική τους υποχρέωση για επιτήρηση και έλεγχο. Επομένω πρέπει να εξετάσουμε τι είδους πληροφορίες συλλέγονταν, για ποιο στόχο, από ποιον και ε, ποιος ήταν ο εντολέας. Και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε μετά από αυτό στην ανάπτυξη μιας συνενετικής συνεργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ένωση μεταξύ των ε, κυβερνήσεων, και πάνω απ' όλα ε, την ανάπτυξη ενός ε, συστήματος δημοκρατικού ελέγχου και εποπτείας του τι γίνεται. Μπορεί λοιπόν η Επιτροπή αυτή να εξετάσει και αν χρειάζεται η τροποποίηση ή οθέτηση συμπληρωματικών πρωτοκόλων στις διάφορες διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις που καλύπτουν τον τομέα αυτών, έτσι ώστε να ενημερωθούν σε σχέση με την εξέλιξη της ε, τεχνολογίας και πρόεδρε αυτή, νομίζω ότι είναι η ουσία των όσων έχει να κάνει η εξαιστική αυτή επιτροπή. Στο συγγνώμη ε, κύριε πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι μέλη της Επιτροπής του Συμβουλίου αλλά θα χρειαστεί να αποχωρήσω γιατί έχω μια άλλη δέσμευση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μποργκέτσι είναι ο τελευταίος στον, στο κατάλογο των ομιλητών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Τα στοιχεία τα οποία εμφανίζονται από τις πρώτες πληροφορίες που είναι αρκετά σημαντικές στον τύπο μας δείχνουν ε, μία εικόνα αρκετά φοβιστική της όλης κατάστασης ότι ε, υπάρχει ένας γενικότερος έλεγχος και μία χειραγώγηση όλων των πληροφοριών που αφορούν ε, τις, τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όταν βλέπουμε ότι αυτό το σύστημα το οποίο ελέγχει όλες τις προφορίες ε, που αφορούν ε, χρηματοπιστωτικές ε, συνδιαλλαγές τα αρχίζουν να δημιουργούνται προβλήματα. Ο καθηγητής ε, Κώστα, ε, ειδικό ε, για τα θέματα λαθρεμπορίου ναρκωτικών, ανέφερε ότι η διακίνηση κεφαλαίων είναι, χρησιμοποιείται για την για να ξεπλύνουμε το μαύρο χρήμα το οποίο χρησιμοποιεί, το οποίο βγαίνει από, την, από το εμπόριο των ναρκωτικών. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε ε, με, μια επιχείρηση αν θέλετε η οποία ε, έχει, η οποία έχει ε, παραβιάσει όλα τα δικαιώματα των πολιτών στο, είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και διαρωτώ με μήπως θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε να εξετάζουμε αυτό το θέμα όπως μας ανέθεσε η Ολομέλεια σαν να είμαστε εμείς μια επιτροπή των, των Ηνωμένων Πολιτειών που έχει την πληροφορία ότι ένας κύριος από, τις, από την Ευρώπη έχει ιδρύει ένα σύστημα που να μπορεί να ελέγχει πληροφορίες που αφορούν όλους τους πολίτες ε, και ε, ξεχνάμε τις διακοπές, ξεχνάμε τα πάντα και ξεκινάμε το έργο μας. Εδώ εμείς ε, θέλουμε να ακούσουμε τον κύριο Σνόουντεν και το λέμε να ακούσουμε, να καλέσουμε και να καλέσουμε ταν Όχι, πρέπει να καλέσουμε και πρέπει να ακούσουμε όλους τους πρωταγωνιστές. Πρέπει να προχωρήσουμε και να ε, καλέσουμε όλους και να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να τους κάνουμε τις ερωτήσεις μας. Θα μπορούσαμε ενδεχόμενα να, και με τηλεδιάσκεψη να μιλήσουμε και με τον ίδιο τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε, διότι αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε τα νόμιμα συμφέροντα αυτών που μας ε, ψήφισαν και τους οποίους εκπροσωπούν. Να πρέπει να ξέρουμε ποιες είναι, ε, ποιος είναι ο σκοπός αυτή του ελέγχου, του παγκόσμιου ελέγχου. Να ξέρουμε ποιες υπερδυνάμεις ε, το την, την ήθελαν, γιατί δεν νομίζω ότι ο πρόεδρος Ομπάμα είναι η πραγματική εξουσία που αποφάσισε όλα αυτά και θα πρέπει να ξέρουμε ε, και τι αρμοδιότητες υπάρχουν. Γιατί θα πρέπει και θα πρέπει να ξέρουμε ε, ποιο μπορεί να ελέγξει κατά πόσον υπάρχουν, α παραδείγματο χάρη, στο, πρόεδρο, στο γραφείο του Προέδρου. Okay, thank you. Σας ευχαριστώ, συνάδελφοι. Δεν ξέρω αν θέλει άλλος κανείς το λόγο. Όχι. Οπότε εκ μέρου του Πρόεδρου Λόπε να κάνω μια ανακεφαλαίωση με τις εξή προτάσεις. Καταρχήν, Ω προ την εντολή. Με βάση ε, το ψήφισμα που εγκρίθηκε στην Ολομέλεια και τη σημερινή συζήτηση, θα πρότεινα στη Γραμματεία να κάνει ένα σχέδιο με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που διατυπώθηκαν προκειμένου να οριστικοποιήσουμε το περιεχόμενο της εντολής και να σας στείλουμε στις επόμενες δύο εβδομάδες ε, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την πρόταση αυτή. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, η Γραμματεία ήδη κατήρτισε ένα κατάλογο με ημερομηνίε για 12 συνεδριάσεις μέχρι τα τέλη του χρόνου. Η πρώτη θα γίνει στις 5 Σεπτεμβρίου το απόγευμα, 3 με 6,5, 7.30 και η δεύτερη μεταξύ 23 και 26 Σεπτεμβρίου θα επιβεβαιωθεί στη συνέχεια. Θα σας στείλουμε και τον κατάλογο με τις προτινόμενες ημερομηνίες για τις συνεδριάσεις. Τρίτον, σε ό,τι αφορά τους ε, καλεσμένους και τους ομιλητές, όλοι όσοι έχουν ε, συγκεκριμένες προτάσεις ε, για προσκεκλημένους να τις στείλουν στη γραμματεία για να συντάξουμε ένα κατάλογο και να δούμε πόσο καιρό έχουμε για να τους στριμώξουμε όλους το πρόγραμμα. Και έχω και μία προσωπική πρόταση, σύσταση. Μετά τις δηλώσεις του Κις Αλεξάνδρερ, του διευθυντή του NSA, ότι ενδιαφέρεται για το διάλογο, θα έλεγα να είναι από τους πρώτους καλεσμένους μας. Ε, και μάλιστα στην Επιτροπή για, το, για τη CIA καλέξαμε τον τότε αρμόδιο του, του τμήματος για την ε, εσωτερική ασφάλεια. Οπότε θα μπορούσαμε κάλλιστα να καλέσουμε τον Διευθυντή της ε, Υπηρεσίας Ασφάλειας ε, των Ηνωμένων Πολιτειών για τον Σεπτέμβριο. Σε ό,τι αφορά τις, ε, την τεκμηρίωση, ενημερωτικά σημειώματα και μελέτες του, του Τμήματος Πολιτικών, καταρχήν μία περιγραφή της κατάστασης, και του εφαρμοστέου δικαίου των ΗΠΑ, το πρόγραμμα Πρίσμα, καθώς και εθνικές νομοθεσίε και εθνικά συστήματα μαζικής παρακολούθησης των κρατών μελών. Να γίνει μια χαρτογράφηση δηλαδή της κατάστασης, να δούμε που έγινε το πρόβλημα. δεύτερο σημείωμα ενημερωτικό, συγκεκριμένη και σαφής ανάλυση για τι συνέχεια δόθηκε στην έκθεση έσελον. Κατά πάσα πιθανότητα αυτό το σημείωμα θα είναι αρκετά συνοπτικό. Τρίτον, σύντομο επίσης ενημερωτικό σημείωμα για το Ίνσεν, δηλαδή ποια είναι η εντολή του, τι ακριβώς κάνουν, τι δεν περιλαμβάνεται στην εντολή, σε ποιον υπόλογη, τι μηχανισμοί εποπτείας, επίβλεψης υπάρχουν και ούτω καθεξής. Τέταρτη πρόταση να ζητήσουμε από τη Γραμματεία να καταρτήσει κατάλογο με σημεία επαφή και στα Εθνικά Κοινοβούλια, ιδιαίτερα σε κοινοβούλια χωρών που γίνονται τέτοιε έρευνε και υπάρχουν τις εξεταστικές επιτροπές, καθώς και ε, με γερουσιαστές που έκαναν ε, δημόσιες δηλώσεις για τέτοια θέματα, ίσω ενδιαφέρονται για συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτέ είναι οι προτάσει μου. Συμφωνείτε? Ο κύριος Σταβάρης. Ένα σύντομο σχόλιο για τα πρακτικά. Να προσκαλέσουμε και τον άνθρωπό μας στη Washington για το πρόγραμμα SWIFT. Γιατί η, η Επιτροπή δεν μας επέτρεψε να τον συναντήσουμε. Μπορεί να έρθει ή να τον καλέσουμε για να δούμε αν υπάρχει διαβίβαση πληροφοριών από το ένα πρόγραμμα στο άλλο. Αυτή τη φορά πιστεύω ότι η Επιτροπή θα πρέπει να μας επιτρέψει να συναντήσουμε αυτόν τον άνθρωπο και κλεισμένο το θυρών εννοείται. Καλώ, συμφωνώ. Αλλά θα ήθελα να ζητήσω από όλε τι ομάδε και του τρει εκπροσώπου τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων να υποβάλουν τι γραπτό τι προτάσει του για καλεσμένου στι ε, ακροάσει. Για να προσπαθήσουμε να τι εντάξουμε στο χρονοδιάγραμμα και να οριστικοποιήσουμε το πρόγραμμα, μέχρι τα τέλη ε, το πρόγραμμα για τα τέλη του έτους. Αν συμφωνείτε λοιπόν, έτσι θα κάνουμε και μπορώ να κηρύξω το πέρα συνεδρίασης. Ευχαριστώ.